Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ο μόνος κανόνας που τηρούμε αυστηρά σε αυτή την Ευρωβουλή είναι ο αυστηρός έλεγχος του χρόνου. Πρέπει να τηρήσω τα 7 λεπτά που μου δίνει η Προεδρία. Και έτσι στην παρέμβασή μου δεν θα μπορέσω να δικαιώσω τις πολλές και εξαιρετικές παρεμβάσεις που έγιναν χθε στην ομάδα εργασίας. Χωρίς να καθυστερήσω θα αρχίσω παρουσιάζοντας τα 7 σημεία που πιστεύω ότι ολοκληρώνουν τα συμπεράσματα αυτής της ομάδας εργασίας. Το πρώτο συμπέρασμα είναι αυτή, ότι αυτή η κρίση, η κρίση που περνάμε, είναι μια κρίση πολύ πιο βαθιά και έντονη, πολύ με μεγαλύτερη εμβέλεια και παγκοσμιοποιημένη μορφή από ό,τι προβλέπαμε. Είναι μια διαρθρωτική κρίση και δεν είναι μια απλή κυκλική κρίση. Η κρίση της 29ης ε, ε, ξεκίνησε στην ΣΥΣΥΠ αλλά κράτησε δύο χρόνια μέχρι να φτάσει στην Ευρώπη του 1929. Η σημερινή κρίση ήταν πολύ ταχύτερη. Μετά την κατάρρευση των Lehman Brothers και της Ισλανδίας ε, δύο εβδομάδες μόνο πέρασαν για να χτυπηθεί να πληγεί η Ευρώπη. Έτσι λοιπόν το συμπέρασμα είναι ότι η θέση της σύνδεσης, δηλαδή ότι οι αναδυόμενες οικονομίες θα μπορούσαν να αναπληγούν, πολύ λιγότερο από ό,τι προβλεπόταν να αναπτύσσεται η Κίνα. Οι οικονομίες της Ρωσίας, Βραζιλίας επίσης υφίστανται τα πλήγματα. Δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι αυτή η δραματική αλλαγή σενάριου προϋποθέτει μια επανάσταση στον τομέα των ιδεών. Μια επανάσταση παρόμοια με εκείνη που έγινε μετά την κρίση του 1929 ή και μετά την κρίση του 1973, την πρώτη πετρελαϊκή κρίση. Πιστεύω τερματίστηκε η ε, περίοδος ε, της ε, χωρίς ρυθμίσεις ανάπτυξης, ξέφρενης ανάπτυξης ή χαλαρών ελέγχων. Και έτσι σε σχέση με την κοινωνική οικονομία της αγοράς, στην οποία αναφέρθηκε και ο πρόεδρος Πέτερινγκ, οικονομία κοινωνική της αγοράς σε σχέση και με τις δημόσιες αρχές και τον καθορισμό κανόνων του παιχνιδιού, ώστε να είναι ο ανταγωνισμός θεμητός και δίκαιος και έτσι να μεριμνήσουμε ώστε η ανάπτυξη θα σέβεται και το περιβάλλον. Τρίτο σημείο. Γίνεται αναφορά εδώ ειδικά στη χρηματοοικονομική κρίση. Όλοι οι παρεμβαίνοντες συμφωνούσαν ότι η αποκατάσταση των χρηματοοικονομικών αγορών πιστοτικών αγορών είναι η αναγκαία εκ των όνων προπόθεση ώστε η αγορά, οι οικονομίες επιχειρήσεις και οικογενειακές επιχειρήσεις να μπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά. Είναι κατεπήγον να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη λοιπόν στα οικονομικά οικονομικά συστήματα. Η νομισματική πολιτική μετά από την τοποθέτηση που δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετική η ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και για τους κανόνες του παιχνιδιού εκφράστηκαν δύο αιτήματα προς τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Μεγαλύτερη ταχύτητα και μεγαλύτερη, μεγαλύτερη τόλμη όσον αφορά τα μέτρα τα οποία θα ε, πρέπει να λυθούν και καθορισμός ε, προθεσμιών μεγαλύτερης διάρκειας χρονικής. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει δύο ανώτατες, έχει ανώτατη περίοδο 6 μηνών, ενώ στην Αμερική υπάρχει περίοδος 3 ετών για την εξόφληση. Έτσι λοιπόν δίνουν, είναι αναγκαίο να υπάρχουν δυνατότητες μακροπρόθεσμης δανειοδότησης και η λειτουργία της διατραπεζικής αγοράς και ο δανεισμός ο διατραπεζικός είναι η δεύτερη προϋπόθεση για να αντιμετωπίσουμε την κρίση μελέτη προϋπόθεση είναι η μείωση των επιτοκίων με τις ενέσεις στις χρηματοπιστωτικές είτε από τα, τις κεντρικές τράπεζες είτε από τα εθνικά συστήματα θα πρέπει να περάσουν το δυνατόν νωρίτερα στις επιχειρήσεις για να είναι λειτουργικές. Η ε, θέσπιση ενός ρυθμιστικού πλαισίου για να υπάρχει διαφάνεια σε σχέση με τα προϊόντα και τους φορείς και τις αγορές και ενίσχυση των μηχανισμών επιτήρησης για να διασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία των χρηματοοικονομικών φορέων είναι η τέταρτη προϋπόθεση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και να ξεπεράσουμε αυτή την ε, χρηματοοικονομική κρίση. Ε, τέλος, μια και είναι παγκοσμιοποιημένη η κρίση και μια είναι και πολύ πιο έντονη η κρίση από ό,τι προβλεπόταν, μια και πλήττει όλο τον κόσμο, μια αναθεώρηση της θεσμοθετημένης αρχιτεκτονικής δομής, δίνοντας μεγαλύτερο πρωταγωνιστικό ρόλο στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στο Financial Stability Forum Τέταρτον, δεν μπορούμε να οπισθοδρομήσουμε σε σχέση με τι προόδου που έχουμε κάνει. Αναφέρομαι στην ενιαία αγορά. Ο ανταγωνισμό πρέπει να λειτουργεί και όσον αφορά τι δημόσιε ενισχύσει σε επιχορηγήσει, καθώ επίση και τι δημόσιε επιδοτήσει στου επιχειρηματικού τομεί και βιομηχανίε που αντιμετωπίζουν δυσκολία. Είναι ένα κεκτημένο που δεν μπορεί να αφήσουμε να υπονομευθεί σε αυτόν τον οικονομικό πόλεμο που ζούμε. Και πέμπτο συμπέρασμα, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε ότι το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη η ισορροπία των δημοσίων οικονομικών είναι μια βασική θεμελιώδης προϋπόθεση για την μακροοικονομική σταθερότητα. Και αυτή η μακροοικονομική σταθερότητα είναι η αναγκαία οικονομική συνθήκη για μια υφόρο ανάπτυξη διαχρονική διάφορες χώρες θα είναι αντικείμενο διαδικασίας επί παραβάση και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθορίσει εκείνα τα σχέδια τα οποία θα επανορθώσουν, θα αποκαταστήσουν τη σημερινή κατάσταση και θα μπορέσουν να δημιουργήσουν μια νέα σταθερή ισορροπία. Έκτο σημείο. Θα ήθελα να αναφερθώ εδώ ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση, δόθηκε έμφαση από τους παρεμβαίνοντες ότι θα πρέπει να συνδυαστούν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα με τα μακροπρόθεσμα μέτρα. Θα υπάρχει ζωή που θα συνεχίζεται και μετά την κρίση. Πρέπει να ξεπεράσουμε λοιπόν αυτή την κρίση με τον καλύτερο τρόπο, όντα περισσότερο ανταγωνιστική και πιο ε, λειτουργική από μέχρι σήμερα. Ε, επισημάθηκε ότι τα τελευταία 20 χρόνια πριν από την κρίση η, οικονομική, ε, η οικονομία τη Ευρώπη σε σχέση με τι οικονομίε των ΗΠΑ και τη Ιαπωνία ε, είχε κάποια απόσταση και ήταν πιο αποτελεσματική σε σχέση με την καταπολέμηση τη παγκοσμιοποίηση τη ΗΠΑ. Για κάθε θέση απασχόληση στις ΕΠΑ ε, δημιουργεί το 1,2 νέες θέσεις ε, σε νέους τομείς ε, στις ΕΠΑ. Για κάθε κατεστραμμένη θέση απασχόλησης σε βιομηχανίες που μετεγκαθίστανται σε αναδυόμενες χώρες, μόνο 0,8 θέσεις απασχόλησης δημιουργούνται. Γι' αυτό πρέπει να επανορθωθούν αυτά τα πράγματα. Με την, το σχέδιο της πολιτικής Λισαβόνας πρέπει να δραστηριοποιηθούμε ώστε να διασφαλίσουμε και να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένη οικονομίας και να αυξήσουμε την παραγωγικότητα. Ιδιαίτερα στον τομέα των υποδομών, εδώ πρέπει να στοχεύσουν τα προγράμματα της Ένωσης, ώστε το πρόγραμμα ανάκαμψης να λειτουργήσει και σε σχέση με το πάγιο κεφάλαιο, ιδιαίτερα εκείνες οι προσπάθειες που θα είναι πιο έντονες και που θα πρέπει να γίνουν για την τεχνολογική πρόοδο και που εδώ θα πρέπει να δώσουμε προσοχή στην ανάπτυξη και στην έρευνα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μεταφραστούν με τον καλύτερο καλύτερο τρόπο, στι καλύτερε διαδικασίε και βελτίωση των προϊόντων, δηλαδή να, οι δαπάνε να μπορέσουν να μεταμορφώσουν αυτήν την νέα δράση. Δεύτερον, ιδιαίτερη προσοχή στι μικρομεσαίε επιχειρήσει, στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, πληροφορία και τεχνολογία. Και σε σχέση με τέτοιου είδου βιομηχανίε που είχαν ακολουθήσει βραδύτερου ρυθμού στην αναδιανομή και στο λιανικό εμπόριο και στην. Ε, ε, αναγκαία συνθήκη να βοηθηθούν οι μικρομεσαίε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ζητήθηκε τελικά η αναθεώρηση όλων των προγραμμάτων των δημοσιονομικών ώστε αυτά να στοχεύουν στις, ε, στους στόχους εκείνους που προανέφερα προηγούμενα. Τελευταίο, έβδομο σημείο, αλλά εξίσου σημαντικό, η αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου. Υπογραμμίστηκε ότι πολλοί από του νόμου και κανόνε, πολλά από τα συστήματα, πολλά από τα ρυθμιστικά πλαίσια που έχουμε ακόμα, ε, ήταν για μια εποχή όπου υπήρχαν ακόμα σύνορα μεταξύ των κρατών η παγκοσμιοποίηση και η κρίση που ήταν μια έκφραση αυτής της παγκοσμιοποίησης δείχνουν ότι πρέπει να αλλάξουμε κατεύθυνση, να αλλάξουμε προσανατολισμό και να προσανατολίσουμε αυτά τα νέα θεσμικά ρυθμιστικά πλαίσια στη νέα πραγματικότητα, η διαφάνεια των αγορών, ιδιαίτερα εκείνων των ε, όπως μεταφορών βιομηχανικών δραστηριοτήτων στο ε, να ολοκληρωθεί η ενιαία εσωτερική αγορά με την οδηγία για τις υπηρεσίες και για τις ε, ε υπηρεσίες για το λιανικό εμπόριο και τις αντίστοιχες η απλούστευση διοικητική για να είναι δυνατή η άμεση ανάπτυξη και δημιουργία συνθήκων για να δρουν ε, σωστά οι επιχειρήσει, επιχειρήσεις, ελαστικότητα τη αγορά εργασία, Εδώ δόθηκε ιδιαίτερη ε, προσοχή στις μορφές flexicurity, ελαστικότητα και ασφάλεια ε, σε σχέση με τι νέε πρωτοβουλίε και από πλευρά τη Προεδρία. Και όλα αυτά να εντάσσονται σε ένα μεγάλο ευρύτερο πλαίσιο, συνεκτικό και συναφές, παγκοσμιοποιημένο, ώστε να μπορέσει η συνθήκη τη. Λισαβόνα ε, να μπορέσει να ε, δώσει μια νέα πρόθεση σε αυτά. Αυτά είναι τα συμπεράσματα, Πρόεδρε, τη ομάδα εργασία. Πολύ ε, εν περιλήψη και πολύ θα έλεγα εν συντομία. Αυτά ήταν τα κυριότερα συμπεράσματα τη ομάδα. Μα Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σα ευχαριστώ. Χωσέ Μανουέλ Γκαρσία Μαργκάλιο. Είσαστε πραγματικά πολύ επικεντρωμένος και με τον καλύτερο τρόπο καλύψατε μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα τα θέματα. Και τώρα περνάμε στην ομάδα εργασίας 2 να δημιουργηθούν θέσει απασχόληση, καταπολέμηση τη φτώχεια, να διασφαλιστεί η ελευθερία τη κυκλοφορία. Ο Λιούμπομιρ Σοντάρεκ, βουλευτή από την Τσεχική Δημοκρατία. Παρακαλώ, συνάδελφε, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Θα προσπαθήσω <clears throat> να συνοψίσω τι συζήτηση μας στη δεύτερη ομάδα εργασίας. Ε, ο τίτλος, το θέμα μας θα είναι οι κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης επειδή πραγματικά οι επιπτώσεις της κρίσης αυτές ε, ε, έχουν αρχίσει να φαίνονται στην πραγματική οικονομία και ξέρουμε ότι σε μικρό χρονικό διάστημα θα αντιμετωπίσουμε αυξημένη ανεργία και κλείσιμο εργοστασίων και αυτό θα επηρεάσει τις τσέπες του κόσμου. Σε όλα τα κράτη-μέλη λαμβάνονται μέτρα για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά με πλήρη σεβασμό της, ε, της αρχής της επικουρικότητας. Όμως ε, γίνεται μεγάλη προσπάθεια για να μην επηρεαστούν αρνητικά οι απασχόληση και οι θέσεις εργασίας. Ακούγονται πολλές ιδέες, πολλές διαφορετικές απόψεις που ε, αποδεικνύουν ότι όλοι έχουν πλήρη συνέστηση της ε, κατάστασης γιατί η κατάσταση φαίνεται να είναι ακόμη πιο σοβαρή επειδή δεν μπορούμε ούτε καν να αξιολογήσουμε και να μετρήσουμε την, ε, την το μέγεθος των τοξικών προϊόντων ή δεν ξέρουμε τι γίνεται ακριβώς με τις ευρωπαϊκές τράπεζες ε, ποια, ποιο είναι το μέγεθος και άρα και η ε, ζημία που θα επιφέρουν αυτά τα τοξικά προϊόντα φοβούμε ότι επειδή ακριβώς δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε σωστά τα πράγματα θα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να περάσουμε σε μια πολύ μακρόχρονη ύφεση είναι περίπλοκο βέβαια να συζητεί κανείς τις κοινωνικές επιπτώσεις ακόμη και αν μιλάει σε πραγματικό χρόνο και έχει συγκεκριμένα στοιχεία. Καταλαβαίνετε ότι υπό αυτές τις συνθήκες που δουλεύουμε τώρα είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως κατά την άποψή μου θα μπορέσει να αντιμετωπίσει το, τα προβλήματα εφόσον αντιδράσει ενωμένα. Γι' αυτό η συνθήκη της Λισαβόνας παίζει ακόμη μεγαλύτερο ρόλο. Μόνο ενωμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που υπάρχουν. Επίσης πρέπει να έχει ισχυρή ηγεσία ε, κατα, ε, στην αντιμετώπιση της και η Λισαβόνα εδώ εξασφαλίζει ε, κάτι τέτοιο. Ε, συζητήσαμε στην ομάδα μας τη στρατηγική της Λισαβόνας και η συνεπής εφαρμογή της ε, αποφασίσαμε όλοι ότι είναι απαραίτητη τα κράτη-μέλη τα οποία ήδη έχουν κάποιες επιτυχίες στην επιτυχία των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση από τα άλλα κράτη-μέλη που δεν έκαναν κάτι αντίστοιχο. Ε, η, είναι, υπάρχουν πολλά άρθρα πολύ σημαντικά στη στρατηγική της Λισαβόνας που θα μπορούσαν να είχαν εφαρμοστεί και θα βοηθούσαν. Αλλά υπάρχει κι άλλο ένα σημαντικό θέμα το οποίο συζητήσαμε, το θέμα της αλληλεγγύης. Πολλοί ζήτησαν ε, ενισχυμένη αλληλεγγύη για τους πιο εκτεθειμένους αν θέλετε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί βλέπουμε οι ανισότητες να μεγαλώνουν και να πλήττονται ιδιαίτερα οι νέοι, οι ηλικιωμένοι και οι ε, πολίτες με χαμηλά εισοδήματα. Η γνώμη η οποία εξεφράστηκε τελικό στην ομάδα μας είναι ότι πρέπει πραγματικά να ε, ε, φροντίσουμε να επιδειξει η κοινωνία μας αλληλεγγύη για, όλους, για όλες αυτές τις ομάδες του πληθυσμού που, που θίγονται ακόμη πιο έντονα και ελέγχθη ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλες οι δυνατότητες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Θα πρέπει τα ταμεία αυτά να είναι τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία που ε, θα χρησιμοποιήσουμε. Ελέγχθη όμως συγχρόνως ότι αυτά τα δύο ταμεία είναι αρκούν. Αρκούν αν θέλετε. Εκείνο το οποίο ίσως χρειάζεται είναι ένα νέο κοινωνικό σύμφωνο. Ένα καινούριο social pact όπως ελέγχθη στην Ευρώπη ε, επίσης έγινε συζήτηση στην ομάδα μας για τις τέσσερις συμπληρωματικές αρχές. Πρώτον είπαμε ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στους πιο θυγόμενους πολίτες, θα πρέπει να φροντίσουμε στην αγορά εργασίας να προσθέσουμε με κατάρτιση και τα ε, ε, προσόντα και ικανότητες. Ε, τρίτον θα πρέπει όπως είπαμε να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά τα χρηματοδοτικά εργαλεία και γι' αυτό το θέμα θα ήθελα να επεκταθώ λιγάκι ε, γιατί επανειλημμένα ε, ε, ε, αναφέρθηκαν τα ευρωομόλογα. Είδαμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες ε, εκδίδουν συνεχώς χρήμα εντός εισαγωγικών και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και η Ευρώπη να κάνει κάτι αντίστοιχο. Αναφέρθηκαν λοιπόν τα Eurobonds, αυτά τα ευρωομόλογα, τα και η χρησιμοποίησή τους και για την αντιμετώπιση ε, των κοινωνικών προβλημάτων και της κοινωνικής αναταραχής αν θέλετε. Ελεγχθεί επίσης ότι ο προστατευτισμός ε, που δεν είναι λόγο είναι η λύση ελέγχθη επανειλημμένα αυτό δεν θα ε, δημιουργήσει θέσει εργασία. Η εσωτερική αγορά είναι το πλαίσιο με στο οποίο πρέπει να κινούμεθα. Ε, και μια και ανέφερα προηγούμενα τις κοινωνικές αναταραχές, συζητήσαμε και το θέμα αυτό, γιατί οι αναταραχές μπορούν να οδηγήσουν σε εθνικισμό, ξενοφοβία ε, και ε, πραγματικά είπαμε ότι η κρίση αυτή δεν είναι απλά οικονομική κρίση είναι κοινωνική κρίση και κρίση των βασικών αξιών ε, στην, εμπλέκονται εδώ όλοι όλες και οι κοινωνικές ελίτ αν θέλετε και γι' αυτό είπαμε ότι η πολιτική διάσταση είναι πάρα πολύ σημαντική και οι πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν πρέπει να είναι διαφανείς και να μπορούν να γίνουν αποδεκτές η Ευρώπη ε, ρισκάρει εδώ το μέλλον της τη μοίρα της, την αντίληψη των πολιτών της ε, είναι σημαντικό να δείξουμε ότι η Ευρώπη είναι αξιόπιστη ε, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα επόμενα χρόνια. Και μια ακόμη παρατήρηση τελική θα ήθελα να κάνω γιατί ξέρω ότι επανελήφθη επανειλημμένος αυτό ότι η συνθήκη της Λισαβόνας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτύχει η Ευρώπη στον αγώνα ε, που ε, δίνουμε στην ναι, χώρα μου στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου θα συζητηθεί σήμερα η συνθήκη της Λισαβόνας και το βράδυ θα γίνει ψηφοφορία. Είμαι πεπισμένος ότι η ψηφοφορία αυτή θα είναι επιτυχής. Ξέρετε λοιπόν ότι ελπίζω λοιπόν ότι η ψηφοφορία μάλλον είμαι πεπισμένος ότι η ψηφοφορία θα τελειώσει ε, σήμερα βρισκόμαστε στο στάδιο ε, ανάλογα με τη διαδικασία ε, βρισκόμαστε στο στάδιο ε, το οποίο θα είναι αποφασιστικό για το μέλλον της Ευρώπης νομίζουμε Πρόεδρος ευχαριστώ πολύ κύριε και για την ε, παρέμβαση και την παρουσίαση αυτό που έγινε χτες στην ομάδα εργασίας και για την αισιοδοξία σας ότι η Τσεχική Βουλή θα υπερψηφίσει τη σύμβαση της ε, Λισαβόνας, τη συνθήκη της Λισαβόνας. Φροντίστε να φύγετε καιρός για να πάτε να ψηφίσετε. Βεβαίω άμα θέλετε μπορείτε να μείνετε. Αλλά τέλος πάντων ε, ας βοηθήσουμε και ας ελπίσουμε ότι η ψηφοφορία θα είναι επιτυχής. Προχωρούμε τώρα στο τρίτο θέμα για τη βιώσιμη Ευρώπη, την οικονομική ανάπτυξη και την, ε, τις αλλαγές του κλίματος. Η κυρία Μπιλιάνα Ηλιέβα Ράεβα είναι η πρώτη ομιλήτρια. Παρακαλώ. mina damer och herrar, i arbetsgrupp 3 ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε η ομάδα 3 έκανε μια αρκετά ζωηρή ε, συζήτηση χτες οφείλω να ομολογήσω υπήρχαν πολλές και διαφορετικές απόψεις αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτό που είπε ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ έχω ε, ε, ονειρεύομαι I have a dream και βεβαίως τα όνειρα είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτή τη στιγμή όταν διατρέχουμε μια σοβαρή οικονομική κρίση και όταν πολλοί από μας ε, φοβούνται ή τρομάζουν σχετικά με το μέλλον. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να δράξουμε αυτή τη μοναδική ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ε, για να αγωνιστούμε ε, να βρούμε μια λύση να βγούμε από το αδιέξοδο της κρίσης αυτής είναι μοναδική ευκαιρία να ε, μελετήσουμε τα πράγματα σε βάθος για να βρούμε τη λύση. Ε, βεβαίως, όπως είπα και προηγουμένως, υπάρχουν φόβοι για το μέλλον, υπάρχουν πολλές αμφιβολίες, ε, ιδιαίτερα σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος και, της την κλιματική αλλαγή. Πολλοί ε, συνάδελφοι είπαν ότι έχουμε, είμαστε υπερβολικά φιλόδεξοι στο παρελθόν και είχαμε πολλές πολλές δώσει πολλές υποσχέσεις όμως εγώ νομίζω ότι αυτό δεν θα πρέπει να μας τρομάζει θα πρέπει να επιδιώξουμε τους στόχους που θέσαμε και να επενδύσουμε αν θέλετε για να φτιάξουμε μια καλή και σωστή Ευρώπη για τα παιδιά μας, για τις επόμενες γενιές. Πρέπει να δούμε επίσης ποιες άλλες δυνατότητες υπάρχουν. υπάρχουν. Ε, υπάρχει τεράστια ανάγκη για επενδύσεις σε τεχνολογίες του περιβάλλοντος. Ε, ε, θα πρέπει στο θέμα αυτό βεβαίως να λάβουμε υπόψη την οικονομική κατάσταση των διαφόρων κρατών μελών δεν μπορούν όλα τα κράτη-μέλη να κάνουν τόσο μεγάλες επενδύσεις αλλά εδώ παίζει σημαντικό ρόλο η έννοια της αλληλεγγύης από εκεί και πέρα υπάρχουν βεβαίως τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία Ευρωπαϊκή Τράπεζα η οποία μπορεί να βοηθήσει για να φτιάξει για να μεταμορφώσουμε τελικά την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια περιβαλλοντική φιλική στο περιβάλλον Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι προσπάθειες αυτές θα βοηθήσουν τον κάθε ένα πολίτη ξεχωριστά και την κοινωνία μας το σύνολό τους Ε, δεν ε, θέλουμε ε, επίσης να παραμείνουμε στην απλή διασύνδεση κάποιων ηλεκτρικών δικτύων παραδείγματος χάρη θέλουμε να αποκτήσει η Ευρώπη και μια κάποια αυτάρκεια μέχρι ενό σημείου αν είναι δυνατόν είδα άλλαξε η κατάσταση στις Ηνωμένε Πολιτείες έχουμε την καινούργια κυβέρνηση Ομπάμα και θα πρέπει να ξεκινήσουμε και να ξεκαθαρίσουμε στην, ε, στους Αμερικανούς ότι και εκείνοι θα πρέπει να κάνουν πράγματα για το περιβάλλον όπως κάνουμε και εμείς. Η... Η σχέση λοιπόν των κλιματικών αλλαγών με τις ευκαιρίες των επενδύσεων σε προϊόντα και τεχνολογίες και ακίνητα αν θέλετε φιλικά προς το περιβάλλον είναι αυτό καινούριο που πρέπει να κάνει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη τα κτίρια που ανέφερα παραδείγματος χάρη είναι ε, που μέχρι τώρα λέγαμε ότι ε, πρέπει να μονώνουμε τις κατοικίες μας και τα κτίρια για να ε, κρατούμε τη θέρμανση στο ιστορικό του κτηρίου τώρα μπορούμε να κάνουμε και το ανάποδο ας πούμε να αφήσουμε τη θερμότητα με καινούργιες τεχνολογίες μόνωσης να βγαίνει από το κτίριο να δημιουργήσουμε λοιπόν μια καλή, ένα καλύτερο περιβάλλον και σίγουρα αυτό θα δημιουργήσει και νέες θέσεις εργασίας εγώ πιστεύω πραγματικά ότι και όλη η ομάδα μου πιστεύει ότι οι περιβαλλοντικές οι επενδύσεις αυτές ε, θα βοηθήσουν, θα φτιάξουν πολλές θέσεις εργασίας. Θα πρέπει να δούμε. Όλα αυτά σημαίνουν ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσπαθήσουν με δημόσια κονδύλια να τονώσουν την ανάπτυξη. Γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε σε μια οικονομική κρίση και αυτά σημαίνουν ότι οι επενδύσεις που έχουν γίνει και θα γίνουν θα πρέπει να είναι οι ευφιέστερες ώστε μακροπρόθεσμα να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Επενδύσεις λοιπόν, επενδύσεις σε άλλες δομές και διαθρώσεις. Για παράδειγμα, για την ενεργειακή αποδοτικότητα, να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση. Στην ομάδα εργασία εχθέ όμω υπογραμμίστηκε επίση ότι είναι σημαντικό να υπάρξει εμπιστοσύνη που θα δημιουργηθεί, πλαίσιο εμπιστοσύνη. Οι ηγετικές, οι δυνάμεις που θα λαμβάνουν αποφάσεις. Βλέπουμε επίσης ότι και στις ΗΠΑ πώς ο Αμερικανικός λαός αισθάνεται ότι έχει τονωθεί, βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση έχει την εντύπωση, ότι υπάρχει ηγεσία, ηγετικός ρόλος από πλευράς των ηγετών που δείχνουν την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί τους σωστούς προσανατολισμούς. Ελπίζω ότι και στην Ευρώπη θα το καταφέρουμε αυτό. Σημαντικό επίσης είναι να καταφέρουμε να πετύχουμε μια κοινή ενεργειακή πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλοί άλλοι το υπογράμμισαν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Στην ίδια κατεύθυνση πρέπει να στοχεύουμε. Έχουμε διαφορετικές ημερήσεις που ενώνονται σε μια κοινή διάταξη εργασιών, ατζέντα, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Τώρα, το ότι τέθηκαν, οι τίθενται στόχοι στο ευρωπαϊκό επίπεδο δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι ικανοποιητικό και ότι επαρκεί. Ε, είναι απόλυτα αναγκαίο κάθε χώρα να αναλάβει τι ευθύνε τη και να συνεχίσει τι προσπάθειε να επιτευχθούν οι στόχοι που θέσαμε ενώπιον μα. Εμεί ε, ω βουλευτέ έχουμε ευθύνε. Πρέπει να συμμετάσχουμε, να συνεργαστούμε, να ευδοκιμήσουν αυτές οι διαδικασίες και οι προσπάθειες. Σημαντικό είναι επίσης και το θέμα της Κοπενχάγης, της συνόδου Κοπενχάγης. Είναι σημαντικό να υπάρξει μια συμφωνία εκεί. Φυσικά δεν μπορούμε να περιοριστούμε σε αυτό το πλαίσιο όταν έχουμε επενδύσεις που θέλουμε να προαγάγουμε. Πρέπει τώρα ήδη αμέσω να ενεργοποιηθούμε και να μην αναμείνουμε άλλο. Γιατί διαφορετικά θα μπορούσε να είναι πολύ πλέον καθυστερημένη οποιαδήποτε δράση. ευφυείς επενδύσεις ε, για τη σωστή αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών με ταυτόχρονη δημιουργία θέσεων απασχόλησης από πλευρά μα. Γνωρίζουμε φυσικά επίσης ότι οι εκπομπές τρύπων είναι παγκοσμιοποιημένο φαινόμενο. Θα πρέπει και στη Ρωσία και στην Κίνα και στην Ινδία να δούμε τι γίνεται και τι θα γίνει. Να προβληματιστούμε, να τους βοηθήσουμε να κάνουν τις σωστές επενδύσει επενδύσεις στη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει σε κάθε χώρα, σε κάθε πολίτη, σε κάθε χώρα να δώσουμε βοήθεια να υπομισθούν οι πολίτες και όλοι τις ευθύνε. Δεν μπορούμε να σταυρώσουμε τα χέρια, να σταυρώσουν άλλοι τα χέρια και να πούμε τι να κάνουμε, δεν υπάρχει λύση για το φαινόμενο των εκπομπών ρήπων. Όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Κάθε ένας πρέπει να υπομισθεί τις ευθύνε του. Εμείς ως βουλευτές πρέπει να προβληματιστούμε και να δούμε πώς έχει η κατάσταση στη χώρα μας και πώς μπορούμε αυτή τη διαδικασία να την δρομολογήσουμε με σωστό τρόπο και να μην αναμείνουμε με χρυσό του αναλάβουν άλλοι, άλλοι άνθρωποι πρωτοβουλίε. Δύο διαφορετικά θέματα αναφέρθηκαν εδώ και τονίστηκαν. Πρόκειται για μια κοινή ενεργειακή αγορά για την δημιουργία τη για την Ευρώπη. Είναι ένα στόχο που πρέπει να προσπαθήσουμε να πετύχουμε προ την κατεύθυνση αυτή. Από βρετανική πλευρά αναφέρθηκε για παράδειγμα ότι ακριβώ η ζήτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργεια αυξάνεται διαρκώ. Και ίσω αυτό θα μπορούσε να είναι μια πορεία προ το μέλλον. Θέλουμε να αποφύγουμε να καταλήξουμε σε μια κατάσταση στην οποία απλά θα αναμένει κανείς ένα υπερδίκτυο να δημιουργηθεί, ένα super grid η Super Network, ένα υπερδίκτυο. Δεν μπορούμε να αναμείνουμε. Μιλήσαμε και για πολλά άλλα θέματα, Πρόεδρε. Το σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να δημιουργηθεί το πλαίσιο για την ε, λειτουργία της ε, διαδικασίας της στρατηγικής της Λισαβόνας και όλα αυτά πρέπει να βαίνουν εκ παραλίλου με την, με την περιβαλλοντική μας πολιτική. Σας ευχαριστώ πολύ για την έκθεσή σας. Θα ήθελα να αναφέρω και στους τρεις εισηγητές και να ευχαριστήσω για τις τρεις καλές εισηγήσεις και να υπενθυμίσω αγαπητοί συνάδελφοι ότι αν θέλετε να υπάρξει παρέμβαση στη γενική συζήτηση και να παρέμβετε θα πρέπει να συμπληρώσετε τα δελτία request for speaking time, έτοιμα για παρέμβαση ως αγορητής. Και τώρα σε σχέση με την ομάδα εργασίας υψηλών αξιωματούχων και πραγματογνωμόνων για τις κλιματικές αλλαγές, παρακαλώ τον συνάδελφο τον κύριο Πρίτανη Άραν Λάρσον. Σας καλωσορίζω θερμά κύριε Άραν Λάρσον και έχετε τον λόγο παρακαλώ. Thank you very much, uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, μέλη των Κοινοβουλίων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε και μπορώ να μιλήσω σε αυτή τη τόσο σημαντική συνάντηση. Θα ήθελα να εστιάσω στην προσοχή μου σε τέσσερις μεγάλες προκλήσεις που κι εσείς σαν ευρωβουλευτές, σαν εθνικοί βουλευτές, σαν άτομα που λαμβάνουν τις αποφάσεις ε, θα πρέπει να, να λάβουν υπόψη. Το ένα είναι να σώσουμε την οικονομία, το δεύτερο είναι να ανορθώσουμε την οικονομία, να επανισορροπήσουμε την οικονομία, το τρίτο ε, και να υπάρχει ε, μια ισορροπία ανάμεσα στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Ασία, ή ε, αποταμιεύσεις, η κατανάλωση και η βιωσιμότητα. Αυτές είναι Αυτές είναι οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσετε και εσείς στην καθημερινή σας ζωή, στην ημερήσια διάταξη, με έναν συντονισμένο και συνεκτικό τρόπο. Η δική μου ε, συνεισφορά θα είναι να, προσφέρω κάποιες, να θέσω κάποιες ερωτήσεις, κάποια θέματα που θα στηρίζονται και στην ε, εμπειρογνωμοσύνη των άλλων. Το βασικότερο είναι να σώσουμε την οικονομία το οικονομικό σύστημα. Το οικονομικό σύστημα ε, εργάζεται αντίθετα από την α, ανοικοδόμηση αν θέλετε της οικονομίας και υπάρχει το θέμα το, το, το, τραπεζικό σύστημα το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας θα πρέπει να, να καθαρίσουμε αν θέλετε τη Wall Street έτσι ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά οι τράπεζες αλλά το νέο πλάνο, το νέο πρόγραμμα των, ε, της προηγούμενης εβδομάδας ε, των 200 δις ε, δολαρίων δεν εντυπωσίασε ούτε τους ειδικούς ούτε τις τράπεζες και τις αγορές. Το πρόγραμμα αυτό αντιμετωπίζει ένα βασικό θέμα, πρόβλημα, την έλλειψη ρευστότητα του συστήματος. Όμως δεν αντιμετωπίζει τα άλλα σοβαρά προβλήματα, τη μαύρη τρύπα, ας πούμε, που είναι ένα γεγονός ένα μεγάλο κομμάτι των ε, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ε, είναι αφαιρέγγια, όπως είπε και ο κύριος Γούλς. Ε, το, το, το δημοσιονομικό σύστημα πρέπει να ξεκαθαρίσει και θα πρέπει όλοι να παίξουμε έναν σημαντικό ρόλο. Οι πολίτες όμως είναι οργισμένοι με τις τράπεζες και οι πολιτικοί δεν μπορούν να παίξουν ε, ένα πολύ μεγάλο ρόλο ε, για την, ε, για την εξυγίαση του τραπεζικού συστήματος. Είναι ένας φαύλος κύκλος, μια κατάσταση κάτσου 22. Ο Στρόσο κάν απίφθινε μια έκκληση έτσι ώστε οι κυβερνήσεις να, να διαρθρώσουν τις τράπεζες, να προσφέρουν δημόσια υποστήριξη, να κλείσει το θέμα των αφαιρέγγιων τραπεζών και να, υπάρχουν νέες, να δημιουργηθούν νέε υπηρεσίες για την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων. Ε, όσον αφορά τώρα τον, την, το regulation, τον, τον διακανονισμό αν θέλετε, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση να δώσει μία λύση έτσι ώστε να δημιουργηθεί μία ε, νέα οικονομική τάξη, το, G, το G20 να επιβληθούν συγκεκριμένοι κανόνες, να είναι σαφείς οι κανόνες λειτουργίας. Ε, εγκρίθηκε την προηγούμενη εβδομάδα ένα, ένα ποσό ε, για ενίσχυση 80 δισεκατομμυρίων ε, ευρώ θα πρέπει να εντυπωσιαστούμε με τα νούμερα αυτά ή θα πρέπει να ε, θεωρήσουμε ότι το βάρος τελικά θα πρέπει να το αναλάβουν οι μελλοντικέ γενιές. Ακούγοντας ε, τις ε, παρουσιάσεις ε, των πολιτικών για την ανάκαμψη της οικονομίας, θα πρέπει να αντιμετωπίσετε με ψυχραιμία τα νούμερα αυτά. Εσείς σαν άτομα τα οποία επιβλέπουν αν θέλετε τις κινήσεις των τραπεζών, των κυβερνήσεων, θα πρέπει να θέσετε κάποιες ερωτήσεις. Παραδείγματο χάρη, ποιες θα πρέπει να είναι, ποιες είναι οι συνέπειες ε, όλων ε, των όσων δεν κάνουν οι κυβερνήσεις ας πούμε και ποιο θα ήταν, ποια θα ήταν η συνέπεια εάν κάνανε κάτι ή πόσο αποτελεσματικά είναι τα μέτρα αυτά για να ε, υπάρχει ενίσχυση της ζήτησης ή όλα αυτά είναι απλώς μια βιτρίνα. Το πρόβλημα είναι δημιουργούμε μια ανταγωνιστική αγορά ή την υποσκάπτουμε. Επίσης Όσον αφορά την μία μόνιμη ανόρθωση της εικονάκαψης της οικονομίας, τι πρέπει να κάνουμε. Τώρα, όσον αφορά τις συνέπειες των μέτρων, θα ήθελα να σας πω ε, αυτά τα οποία είπε ο καθηγητής του Στάνφορντ, ο κύριος Πέντς, ο οποίος ήταν και Νόμπελ ε, το 2001, είπε ότι η κρίση ξεκίνησε στον ε, οικονομικό τομέα και ο οικονομικός τομέας είναι πάρα πολύ σημαντικός όταν θέλουμε να βρούμε κάποιες συγκεκριμένες λύσεις και όχι όταν θέλουμε να σώσουμε τις τράπεζες και λέει ο κύριος Στένς, δεν θέλουμε απλώς ένα πακέτο ενθάρρυνσης, αλλά θέλουμε μια, ένα πιο συστηματικό πρόγραμμα δημιουργίας περιουσιακών στοιχείων και νομίζω ότι τα θέματα των δανείων όσον αφορά την αγορά σπιτιών θα είναι, θα είναι μια πάρα πολύ καλή αφιτηρία. Αυτό, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις Ηνωμένε Πολιτείες. Και οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκράτες θέλουν να βρουν τρόπους για να λύσουν το θέμα αυτό, το, το, οικοδομικό και τον, το στεγαστικό και ίσω υπάρχουν και κάποια προβλήματα και στην Ευρώπη. Τώρα, να κάνω κάποια σχόλια όσον αφορά την κοινωνική πολιτική, που είναι αναπόσπαστο τμήμα για την ανόρθωση της οικονομίας. Οι κοινωνικέ πολιτικές θα πρέπει να αποτελέσουν μια προϋπόθεση και όχι μια πολυτέλεια την οποία μπορούμε να ανεχτούμε μόνο στα καλά χρόνια. Οι ορισμένες χώρες όμως η κοινωνική πολιτική δεν χρηματοδοτείται επαρκώς και δεν μπορεί να αντισταθμίσει την μείωση της ζήτησης. Και εάν είχαμε ένα καλύτερο σύστημα επιδοτήσεων, ίσως να ήταν και καλύτερες οι συνέπειες και για τις τράπεζες. Αυτά, δεν τα, αυτά τα λένε και οι Financial Times ούτως ή άλλως. Συμφωνώ απόλυτα με τους Financial Times. Η κοινωνική πολιτική θα μας δημιουργήσει ένα καλύτερο τραπεζικό σύστημα για το μέλλον. Τώρα, για να, πώς θα μπορούσαμε να σώσουμε το χρηματοπιστωτικό σύστημα και να ανορθωθεί η οικονομία. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών πληρωμών στις, στις Ηνωμένε Πολιτείε είναι πάρα πολύ ψηλό. Το ίδιο είναι και στην Κίνα και στην Ιαπωνία και σε όλη την Ανατολική Ασία. Αυτό είναι ένα έλλειμμα το οποίο δεν μπορεί να παραμείνει. Δεν μπορούμε να ε, στηριχθούμε σε ένα ε, μακροοικονομικό ασταθές σύστημα. Η Ευρώπη πρέπει να ε, περιμένει μάλλον τώρα, κρατώντας μια αμυντική στάση και περιμένει τους άλλους κάτι να κάνουν. Η Ευρώπη όμως πρέπει να χρησιμοποιήσει τη δύναμή της, τη δύναμή της σαν, ένα, σαν μια δύναμη ομαδική και Βέβαια, προφανώς οι προστατευτικές κινήσεις υποσκάπτουν ε, και, το, και τις αγορές αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Πέραν όλων αυτών των προκλήσεων όμως, τις οποίες εσείς αντιμετωπίζετε, υπάρχει και μια τέταρτη πρόκληση που είναι την, η αναδιάρθρωση του όλου ενεργειακού συστήματος και αυτή είναι μια αυτόνομη πρόκληση και κάποιο κεφάλαιο σε όλα τα συστήματα ανάκαμψης. Ε, λαμβάνοντας υπόψη είναι την ανάλυση του Νίκολα Στέρνς για τις κλιματολογικές αλλαγές, είπε ότι η, η στρατηγική για το κλίμα είναι η ε, πλέον σωστή στρατηγική που μπορούμε να ακολουθήσουμε και οι επενδύσεις στον πυρηνικό τομέα είναι σημαντικές έχει ένα καλό, ε, με καλό αντίκτυπο, ανθερθητικό αντίκτυπο και στις επενδύσεις αλλά και στην πίστη των καταναλωτών, των επενδυτών. Και θα πρέπει να προσθέσω μία σύσταση όσον αφορά τις διαδικασίες ε, των ε, ευρωπαϊκών πολιτικών στα τελευταία δέκα χρόνια δημιουργήσαμε δύο μεγάλες ε, στρατηγικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Λισαβόνα για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την στρατηγική για την ε, βιώσιμη ανάπτυξη και τώρα έχουμε και μια τρίτη την στρατηγική για την ανόρθωση, για την ανάκαμψη για να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη. Αυτές θα επικαλύπτονται οι στρατηγικές και θα προσπαθήσουν να μονοπολίσουν την ε, θέληση και, τις, ε, και την χρηματοδότηση των πολιτικών. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας συντονισμός ανάμεσα σε αυτές τις τρεις στρατηγικές. Επίσης, να σας πω και μια ιδέα μου για το πόσο θα κρατήσει ε, αυτή η κρίση και πόσο βαθιά θα είναι αυτή η κρίση. Ένας από αυτούς που προέβλεπε αυτή την, την κρίση ήταν ένας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, ο Νοριέκ ο και α δούμε τι πιστεύει για το μέλλον αυτό ο άνθρωπο. Σε μια συνέντευξη που έδωσε πριν από μερικέ μέρες, είπε ότι η παρούσα κρίση θα είναι τρεις φορές πιο βαθιά και, τρεις, και θα κρατήσει τρει φορέ περισσότερο από την τελευταία κρίση. Λαμβάνοντα υπόψη όμω ότι θα κάνουμε όλε τι κινήσεις μας σωστά, προσπαθώντας να σώσουμε τις τράπεζες και να ανακάμψουμε την οικονομία. Βέβαια, τον υπογραμμίζω αυτό, αρκεί να κάνουμε όλες τις σωστές κινήσεις όσον αφορά την δημόσια ε, πολιτική. Και σα εύχομαι κάθε τύχη να, να πάρετε τις σωστές αποφάσεις σε αυτούς τους δύσκολους κερνούς που περνάμε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ καθηγητά Λάρσον για τη δήλωσή σας, τοποθέτησή σας. Χρειαζόμαστε καλές συμβουλές ώστε οι πολιτικοί να κάνουν τα σωστά πράγματα. Και πάλι σας ευχαριστούμε. Και τώρα θα δώσω την πρωτοκαθεδρία στον Προεδρεύοντα Πρόεδρο κύριο Σομπότκα παρακαλώ. Ευχαριστώ. κύριε και κύριοι, θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας που είχαμε ξεκινήσει χθε, θα την συνεχίσουμε τώρα εδώ. Θα ήθελα όλους να τους παρακαλέσω να τηρήσουν τα δύο λεπτά ως όριο για τις παρεμβάσεις. Ο κύριος ε, Λατούσας από την Λιθουανική ΣΕΙΜ, από τη Λιθουανική Βουλή. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι ακούσαμε πολλές καλές συμβουλές ε, αυτές ε, τις ημέρες και χθε και σήμερα. Τα συμπεράσματα των ομάδων εργασιών είναι βέβαια και αυτά πολύ ενδιαφέροντα. Θα ήθελα να επανέλθω σε ένα επίκαιρο θέμα και να πω ότι καλωσορίζω την απόφαση να υπάρξουν νέα κονδύλια που θα διατεθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μέρο αυτών των κονδυλίων να χρησιμοποιηθούν για ενεργειακά προγράμματα. Η κρίση φυσικού αερίου κατέδειξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ιδιαίτερα ευάλωτη, επειδή εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από μονοπόλια στον ανεφοδιασμό ενεργειακών προϊόντων τη. Και όλοι θα συμφωνούσαν σήμερα ότι η ενεργειακή διασφάλιση θα έπρεπε να είναι εξασφάλιση πάνω πάνω στην ημερήσια διάταξη. Και τώρα για αυτά τα ε, ποσά και ένα μεγάλο μέρος αυτού που θα πρέπει να στραφούν στα ενεργειακά προγράμματα είναι μια πολύ έγκαιρη απάντηση και αντίδραση στην ε, δεδομένη αυτή κατάσταση έντονης ανάγκης. Και αναλογικά σε σχέση με τα όσα έχουμε διαθέσιμα θα πρέπει έτσι να δράσουμε. Αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό για χώρες που έχουν αποκοπεί, ε, δεν βρίσκονται εντεταγμένες στην ευρωπαϊκή αγορά Ενεργεια και θα βοηθήσει να ξεπεράσουν αυτές οι χώρες και τις οικονομικές δυσκολίες ο παρόν προπολογισμό δεν έχει άλλη εναλλακτική λύση από το να χρησιμοποιήσει κάποιο πλαίσιο ελαστικότητα και να προκαθορίσει κάποια κονδύλια για αυτή τη χρήση. Είναι νομίζω μια σωστή αντίδραση αυτή. Κατανοώ βέβαια από την άλλη πλευρά το θέμα της ε, δημοσιονομικής ε, ευελιξίας θα συζητηθεί μέσα στο πλαίσιο της δημοσιονομικής αναθεώρησης. Όμως αυτά τα θέματα θα πρέπει τώρα να αντιμετωπιστούν. Η πρόσφατη κρίση φυσικού αερίου καταδεικνύει τον κατεπήγοντα χαρακτήρα αυτή τη δράση. Η Λιθουανία και οι χώρε τη Βαλτική θα αντιμετωπίσουν ένα χωρί προηγούμενο πρόβλημα ενεργειακού ανεφοδιασμού, ιδιαίτερα μετά το κλείσιμο Λιθουανία του πυρηνικού αντιδραστήρα της Σιγναλίνα. Και δείχνουμε κάθε κατανόηση και κατανοούμε τα προβλήματα των χωρών που υφίστανται πλήγματα από την κρίση φυσικού αερίου. Αν είχε κρατήσει επί μεγαλύτερο διάστημα αυτή η κρίση φυσικού αερίου, δεν μπορώ να φανταστώ πώ οι κυβερνήσει αυτών των χωρών θα μπορούσαν να επεξηγήσουν στου πολίτε του το ότι δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τι ε, εντόπιες δυνατότητες δεδομένης και της μη διασύνδεσής τους με το δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας έχει τεράστια σημασία για αυτές τις χώρες. Απευθύνω έκκληση στο ΕΚΟΦΗΝ, στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Επιτροπή Προϋπολογισμών να κάνουν κάθε προσπάθεια για τη συμφωνία, επίτευξη συμφωνίας για τη διάθεση αυτών των κονδυλίων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Στη συνέχεια Λούτζεκ Σέφτικ από την Τσεχική Γερουσία. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να πω ότι έχω πείρα σε σχέση με διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις και διασκέψεις όσον αφορά και το Ευρωκοινοβούλιο και τη συμμετοχή του και την, ε, το έργο της ε, ομάδας ε, WinCock είχαμε και πολύ χρήσιμα συμπεράσματα και συναντήσεις με την Ευρωβουλή στο θέμα της ανταγωνιστικότητας για παράδειγμα. Θα έλεγα λοιπόν η ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορέσει να λειτουργήσει σωστά αν βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Αυτός θα είναι ο πύχης, ο γνώμονας με τον οποίο θα μετρηθούν όλα. Θα ήθελα να πω ότι υπάρχει ανάγκη αλλαγή των συμπερασμάτων. Παρόλη την χρηματοπιστωτική κρίση, την τραπεζική κρίση που μετετράπησε μια οικονομική κρίση, δεν θα έπρεπε να αλλοιώσουμε τα συμπεράσματα στα οποία είχαμε καταλήξει στην χθεσινή μας συνεδρίαση, συνδιάσκεψη κάθετα απορρίψαμε τον προστατευτισμό. Όλες οι ομάδες εργασίας και όλες οι κοινοβουλευτικές πολιτικές ομάδες το υπεγράμμισαν αυτό. Πρέπει να καταπολεμηθεί ο προστατευτισμός. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να θυμόμαστε και σε σχέση με κάθε εκλογή. Όχι μόνο για τις ευρωεκλογές αλλά και για τις εθνικές εκλογές στα κράτη-μέλη. Τούτων λεχθέντων ο προστατευτισμός και τα προσκόμματα και οι φραγμοί δεν είναι κάτι που υφίσταται μεταξύ χωρών μόνο, αλλά κάποιοι λομπιίστες προσπαθούν να αποκομίσουν ωφέλη και κέρδος για τους δικούς τους πελάτες και αυτό είναι κάτι που πρέπει κάθετα να απορρίψουμε και θα πρέπει να συνεργαστούμε όλοι από κοινού για μια ενεργειακή πολιτική στην Ευρώπη, ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση με τον πιο επιτυχή τρόπο. Διότι <clears throat> αν δεν μας σκοτώσει θα πρέπει να μας δυναμώσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ναι, ο Πρόεδρος τώρα από την Ευρωβουλή θα παρέμβει ο κύριος Βοτσεχόφσκι. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε μάλλον τα όσα εμφανίστηκαν στο website για την σημερινή συνεδρίαση και για τα συμπεράσματα των ομάδων θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά και ε, δείχνουν ακριβώς ε, τι πιστεύουμε και θα πρέπει να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Η, κρίση, η παγκόσμια οικονομική κρίση δείχνει ακριβώς ε, πώς λειτουργεί ένα ντόμινο και βλέπουμε όμως ότι οι λόγοι για την επιβράδυνση των οικονομιών διαφέρουν. Η Πολωνία έχει την δυνατότητα να τα πάει καλά. Τα τελευταία στοιχεία όσον αφορά τους διάφορους δείκτες που υπολόγισε ο ΣΑ δείχνουν ότι στο τρίτο το τρίμηνο αυτούς τους, αυτής της, χώρα, της ε, χρονιάς θα ανακάμψει η οικονομία μας. Κάθε χώρα έχει αντιμετωπίσει διαφορετικά προβλήματα. Στην Πολωνία το εργατικό κόστος είναι πάρα πολύ υψηλό. Θα ήταν καλό εάν είχαμε ε, βελτιωμένους μηχανισμούς επίβλεψης και επιθεώρησης, ε, όπως επίσης και αν η κυβέρνηση ασχολείται για να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις με πιο γρήγορο ρυθμό. Το Εθνικό Κοινοβούλιο της Πολωνίας ε, πήρε μέρος στην συζήτησή μας και ε, θα ήθελα να επιστρέψω την προσοχή σας σε ένα άλλο στοιχείο. Το οικονομικό πρόγραμμα ανάκαμψης ε, αναφέρεται στο πώς θα μπορούσε να ξεκινήσει μια δουλειά οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε τρεις μέρες χωρίς κόστος. Αυτό όμως το startup, το μηχανισμό startup ε, μιας εταιρείας δεν λειτουργεί στην χώρα μου. Επομένως οι υπηρεσίες ε, που προσφέρονται από την, ε, από το δημόσιο δεν, μπορεί, δεν είναι αποτελεσματικές, δεν έχουν καμία συνέπεια. Για να ξεκινήσει μια εταιρεία στην επιχείρηση στην Πολωνία χρειάζεται 30 μέρες και 700 ε, ευρώ που είναι πολύ πιο υψηλό ποσό σε σχέση με τα όσα ισχύουν στην, στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν θα, μπορούσαμε να, θα μπορούσε κανείς να βοηθήσει ε, ε κάποιος ξένος την κατάσταση στην Πολωνία. Όχι βέβαια, διότι δεν έχει καμία ε, αρμοδιότητα. Και ελπίζω ότι θα αλλάξει αυτό και πιστεύω ότι αυτό θα είναι ένα μικρό βήμα για, μια, για ένα νέο οικονομικό deal στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λόγο τον έχει τώρα από το Σουηδικό Κοινοβούλιο η κυρία Καρίνα Άντολφσον Έλγκεστάμα. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και θα ήθελα εγώ να αναφερθώ στην στρατηγική της Λισαβόνας και πρόκειται για το μέλλον αυτής της στρατηγικής Λισαβόνας. Αυτό που βλέπουμε σήμερα ήδη και πολλοί το προανέφεραν είναι το ότι βρισκόμαστε σε μια χρηματοοικονομική κρίση. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι οι οικονομικές αγορές ξεπέρασαν τις δυνατότητές τους και αντιμετωπίζουν τώρα προβλήματα. Και αυτό πλήττει όλο τον πληθυσμό. Οδηγεί σε μεγάλη ανεργία, οδηγεί σε ενισχυμένα έντονα, κοινωνικά, ε, ιδιαίτερα έντονα κοινωνικά προβλήματα. Και βλέπουμε ότι όχι μόνο έχασαν τις θέσεις απασχόλησης ε, πολίτες, αλλά έχασαν και τα σπίτια τους. Και θα έλεγα αυτό που ο συνάδελφος χθε από πλευρά της Ευρωβουλής είχε αναφέρει μπορεί πλήρως να υποστηριχθεί και από μένα. Το μέλλον της στρατηγικής λοιπόν τη Λισαβόνα είναι σημαντικό. Πρέπει να είναι όμως μια στρατηγική που θα ενισχύει περισσότερο την ανθρώπινη συνιστόσα, την συνιστόσα των πολιτών στην ανθρώπινη πτυχή τους. Και αυτό όχι επειδή μια κοινωνική πολιτική θα πρέπει να ακολουθεί, αλλά επειδή η κοινωνική πολιτική θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ω παραγωγικό τομέα, Πρόκειται για το θέμα των ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων. Η στρατηγική της Λισαβόνας θα πρέπει να είναι μια στρατηγική όπου σε όλους τους τομείς τα ίσα δικαιώματα και η ισότιμη συμμετοχή, ίδιες ίσες ευκαιρίες και ίδια δικαιώματα για άνδρες και γυναίκες θα πρέπει να ισχύουν. Ίδιες προϋποθέσεις και όροι για την ίδρυση μιας επιχείρησης και τη λειτουργία της. Υπό τους ίδιους ε, όρους και προϋποθέσεις του παιχνιδιού. Αυτό είναι τεράστια σημασία αν θέλουμε να δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνη για το μέλλον. Και αν θέλουμε να το καταφέρουμε στο μέλλον να κάνουμε περισσότερα για την απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Το eh, ευχαριστώ. Η κυρία Γιάννα Μπομποσίκοβα, Ευρωβουλευτή, παρακαλώ, θα λάβει τον λόγο. Δεν παρίσταται όμω. Τότε λοιπόν, ο επόμενο αγορητή, Μάκομ ε, Χάρμπορ, Ευρωβουλευτή, παρακαλώ. Uh, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν ε, βλέπω το όνομά μου στο κατάλογο, αλλά τέλο πάντων δεν πειράζει. Εγώ θα μιλήσω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λάρσον, ε, τον καθηγητή Λάρσον για την παρουσίασή του. Είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε ε, τις προκλήσεις που υπάρχουν για όλους μας και είναι πολύ σημαντικός και ο τίτλος της συνάντησης εδώ που λέει New Deal Υπάρχουν πολλές προκλήσεις, υπάρχουν προβλήματα λόγου χάρη στον ε, τομέα των ακινήτων, της στέγασης και ελέγχθησαν πολλά πράγματα στην ομάδα εργασίας ε, όπως ακούσαμε πριν για την ενέργεια, την αποδοτικότητα των κτηρίων, τα καινούργια κτίρια ε, που πρέπει να έχει η Ευρώπη αν θέλει να αντιμετωπίσει και τις κλιματικές αλλαγές. Είναι σημαντικά όλα αυτά. Το καινούριο deal θα πρέπει να περιλαμβάνει και τέτοιες πτυχές ε, και για τα κίνητα και για την, τις και συνδέσεις και για την ενέργεια και τα ενεργειακά δίκτυα κτλ. Όταν μιλάμε λοιπόν για New Deal θα πρέπει να μιλούμε και για αυτά τα πράγματα και όχι μόνο για το πώς θα αλλάξει η φορολογία. Αλλιώς μιλάμε για ένα New Deal που ε, σχεδιάστηκε από μια Αμερικανική κυβέρνηση πριν από δεν ξέρω πόσα χρόνια. Ή, ακούστηκε επίσης ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα η μαύρη τρύπα ελέγχθηκε αυτό χτες σε μια ομάδα εργασίας οι, πρόσ, οι πρόσφατες υφέσεις στις Ευρώπης στις πρόσφατες υφέσεις τι έγινε οι τράπεζες κατάφεραν να ξεπεράσουν τα προβλήματα για πρώτη φορά όμως ζούμε μια ύφεση όπου οι τράπεζες δημιούργησαν τα προβλήματα πρόκειται για κάτι πρωτόγνωρο λοιπόν ο κ. Λάρσον είπε λοιπόν ότι πρέπει να δούμε καινούργιες λύσεις, από καινούργιες οπτικές γωνίες. Η μαύρη τρύπα μπορεί να καλυφθεί ε, από δημ, δημόσιες δράσεις αν θέλετε ή μήπως ε, υπάρχει, υπάρχουν, υπάρχει αδιαφάνεια και κάποια προβλήματα ε, στη, στους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή εταιριών είναι προβλήματα τα οποία μπορούν να ξεπεραστούν προσωρινά και θα ξαναρθούμε σε μια καλύτερη κατάσταση στο μέλλον. Δεν τα ξέρουμε όλα αυτά. Το, και, το New Deal πάντως για μένα, για την άποψή μου είναι παρέμβαση του δημοσίου, των δημοσίων οικονομικών αλλά και προσπάθεια να ξεπεραστεί η μαύρη τρύπα η οποία μαύρη τρύπα είναι όντως άγνωστη Ευχαριστώ και εγώ ευχαριστώ λέει ο πρόεδρος θα ήθελα να τηρήσετε το χρόνο αγόρευσης όλοι μας προχωρούμε στον κύριο Πανιό από τη Γαλλία Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να χαιρετήσω ε, και να ευχαριστήσω για την οργάνωση αυτής της συνάντησης ανάμεσα στους ευρωβουλευτές και στους εθνικούς βουλευτές και να χαιρετήσω και τα συμπεράσματα των τριών ομάδων εργασίας ε, τα οποία μας παρουσιάστηκαν σήμερα το πρωί. Θα ήθελα να εκφράσω τρεις θελήσεις. Το ένα είναι να απευθύνουμε μια έκκληση για να ξεκινήσουν πολιτικές ανάκαμψεις σε όλες τις χώρες. Δεύτερον, να μην περιοριστούμε μόνο στα άμεσα μέτρα για, την, για να ξεφύγουμε από την κρίση, αλλά να υιοθετήσουμε όλα τα μέτρα συντονισμένα για, ε, μεσοπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα για να έχουμε ανταγωνιστικότητα, βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων απασχόλησης ε, και να αντιμετωπίσουμε τι παγκόσμιε προκλήσει. Τρίτον, ε, είναι να μην επανέλθουμε στον προστατευτισμό και μια και είμαστε εδώ και συζητάμε μεταξύ μας, να σας πω ότι κάποιες αποφάσεις που λαμβάνονται προσωρινά για την ε, ενίσχυση κάποιας, κάποιου βιομηχανικού κλάδου, παραδείγματος χάρη το βιομηχανία στην ε, Ευρώπη, ε, θα διατηρηθούν, είναι δεν θα επηρεάσουν άλλες χώρες, γιατί μιλάμε για, μια, για προσωρινά μέτρα συντήρησης και όντως θα πρέπει να υπάρχει ένας διάλογος συντονισμένος έτσι ώστε να επωφεληθούμε όλες οι ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν και στη διαδικασία της Λισαβόνας να έχουμε μια ε, Ευρώπη ε, αποτελεσματική, ε, δραστήρια για να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση, της, να, λειτουργεί και να ενεργεί υπέρ της κοινωνικής πολιτικής και κατά της θέρμανσης του, του πλανήτη μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει ο πρόεδρος, ο επόμενος ομιλητής είναι από την Κύπρο, ο κύριος ε, Παπαδόπουλος. Α, όχι, όχι. Ο κύριος Παπαδόπουλος είναι παρόν, στην αίθουσα. Εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Προεδρείο για την εγγραφή αυτού του θέματος και ιδιαίτερα τις ε, τρεις επιτροπές που έχουν καταλήξει στα συμπεράσματα που μας έχουν ε, παραδώσει. Για να μην επαναλαμβάνω πολλά από τα θέματα που έχουν ήδη ε, αναφερθεί, συμφωνώ και εγώ ότι χρειαζόμαστε μια σειρά μέτρων που θα βγάλει την Ευρώπη από αυτήν την οικονομική κρίση. Θεωρώ ότι έχουμε ήδη καθυστερήσει στην λήψη μέτρων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μια πρέπει να μιλήσουν ε, δύο ε, ε, εθνικοί βουλευτές και μετά ένας ευρωβουλευτής. Ο κύριος Μπούλμαν έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Συμφωνώ με αυτού που μίλησαν για την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Όντω, η ανταγωνιστικότητα ήταν και είναι σημαντική στα πλαίσια τη στρατηγική τη Λισαβόνα. Σωστό. Αλλά αλλά βρισκόμαστε στην κρίση που βρισκόμαστε επειδή δεν είμαστε ανταγωνιστικοί, όχι σε σχέση με αυτά που γίνονταν τα παλιότερα χρόνια βεβαίως έχουν αλλάξει πράγματα στην Ευρώπη αλλά η κρίση προέρχεται από τον χρηματοπιστωτικό πονέα όπου δεν υπήρχαν αυστηροί κανόνες όπου υπήρξε κερδοσκοπία και η κρίση αυτή του χρηματοπιστωτικού τομέα επηρεάζει τώρα την πραγματική οικονομία αυτό το, ε, αυτό το πρόβλημα πρέπει να λύσουμε και θα ήθελα να υπενθυμίσω σχετικά ότι η Κομισιόν υποσχέθηκε να ε, επιδιώξει στόχους και αποτελέσματα του G20 και να κάνει συγκεκριμένες προτάσεις, να αναλάβει πρωτοβουλίες και τελπά. Συγγνώμη, περιμένουμε ακόμη όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που πρόκειται να πάρει η Κομισιόν και που λέγονταν στην έκθεση Λένε και Ρασμούσεν, αλλά τίποτα δεν έχει γίνει. Η χρηματοπιστωτική αγορά λόγω της το ότι μιλάμε για αυτή την αγορά η, απαιτεί την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κάνει τίποτα. Τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας δεν είναι παρκή για να αντιμετωπίσουμε την κρίση, για να μπορέσουμε να ε, αγωνιστούμε όπως πρέπει. Καλύτερο συντονισμός χρειάζεται, εξυγχρονισμός χρειάζεται, καλύτερες επενδύσεις στη διάφορα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τον κόσμο από την πλευρά των εσόδων, των εισοδημάτων. Αυτά είναι αυτά που πρέπει να κάνουμε και πρέπει παντού και και στα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να φροντίσουμε να γίνουν αυτές οι βελτιωτικές αλλαγές. Ευχαριστώ πολύ λέει ο πρόεδρος Ντανιέλ Γκαρίγκ από, το, από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, τρει παρατηρήσει να κάνω. Καταρχά, να χαιρετήσω το ρόλο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διότι όταν αντιμετωπίσαμε τι πιο δύσκολε στιγμέ τη κρίση, είμαστε στο, στην χαράδρα, είμαστε έτοιμοι να επιδείξουμε. Ε, όταν είδαμε τι έγινε στην Αμερική με, τις, ε, με την Lehman Brothers, ε, θα πρέπει να χαρούμε ε, για την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία έδρασε άμεσα και αποτελεσματικό. Ε, θα πρέπει να σας πω ότι συμφωνούμε απόλυτα με την Ευρώπη χωρίς σύνορα, κυρίως στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως θα ήθελα να πω επίσης ότι αντί να έχουμε ένα New Deal υπάρχει, υπάρχουν δύο άλλες έννοιες ή δύο άλλες θεωρίες που επικρατούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή και που θα πρέπει να αναπτυχθούν κατά την άποψή μας. Καταρχάς η κοινωνική οικονομία της αγοράς. Αυτό είναι κάτι στο οποίο αναφέρονται πολλά κείμενα και η συνθήκη της Λισαβόνας αναφέρεται σε αυτό. Δεν μιλάμε απλώς και μόνο για μια απόλυτη ελεύθερη ανταλλαγή, αλλά μιλάμε μιλάμε για μια αγορά την οποία δεν την υφιστάμεθα αλλά την ελέγχουμε και εκεί μπορούν να εφαρμοστούν διάφορες έννοιες σαν και αυτές που ανέπτυξαν οι Ιδανοί συνάδελφοι με την Flexi Security. Επίσης μια άλλη θεωρία είναι η στρατηγική. Έχουμε τη στρατηγική της Λισαβόνας η οποία όμως είναι αδύναμη διότι ε, ε, ε, εξαρτάται από την καλή θέληση των διαφόρων κρατών. Και αυτό το οποίο χρειάζεται τώρα η Ευρώπη να έχει μια πραγματική, μια ουσιαστική στρατηγική, κυρίω στον τομέα τη έρευνα, να έχει μια πολιτική έρευνα που να είναι πολύ πιο ολοκληρωμένη μέσα στα, πλαίσια των προγραμ... μέσα στα προγράμματα πλαίσια δεν υπάρχει συντονισμό αυτή τη στιγμή. Επίση ε, για τη βιομηχανική πολιτική όλοι μιλάνε για τη βιομηχανική πολιτική. Άλλοι λένε, ε, ε την αναφέρουν ανοιχτά, άλλοι θεωρούν, ε, αναφέρονται σε αυτήν έμεσα. όμω αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι μια, μια ουσιαστική βιομηχανική πολιτική, την οποία να τη θέλει η Ευρώπη. Και από την άλλη πλευρά θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει ικανότητε ανάλυση και αντίδραση στου διεθνεί ανταγωνιστέ μα, διότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλους αυτούς ε, τους ανταγωνιστές που μας περιβάλλουν. Ε, χρειαζόμαστε, ε, χρειαζόμαστε κάποια εργαλεία, κάποια μέτρα όταν αντιμετωπίζουμε ας πούμε, έναν αθέμητο ανταγωνισμό. Δεν είναι προστατευτισμός αυτός. Χρειαζόμαστε κάποια ουσιαστικά μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ο επόμενος ομιλητής από την Πολωνική Γερουσία, ο κύριος Μούλοβιτς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, η συζήτηση σήμερα και χθες ήταν χρήσιμη σίγουρα και ήταν και πολύ σχηδής. Η ίδια η κρίση τώρα είναι ιδιαίτερα περίπλοκο φαινόμενο, σύνθετο φαινόμενο το εκτιμώ το ότι βρίσκομαι εδώ και μου δίνεται η δυνατότητα να παραστώ ως μέλος ε, της ε, Επιτροπής Οικονομικών Νομισματικών Υποθέσεων στην Πολωνική Γερουσία και μπορώ να συμμετάσχω. Θέλω να υπογραμμίσω ότι μόνο συντονισμένη δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο κρατών μελών μπορεί να πετύχει τα αποτελέσματα τα οποία ζητούμε και θέλουμε να επιτευχθούν. Από την άλλη πλευρά, η κρίση αποτελεί επίσης και μια ευκαιρία που μας προσφέρεται και αυτό ιδιαίτερα σε εκείνους τους τομείς όπου η Ευρώπη χωλαίνει και βρίσκεται πίσω από άλλες οικονομίες, όπως στον τομέα της έρευνας. Θα απαιτήσει λοιπόν συνεργασία και συντονισμό να καλύψουμε αυτή την απόσταση συνεργασία και συντονισμό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απάντηση στην κρίση βρίσκεται, έγκυται στην ίδια την ε, οικονομία και το πνεύμα του επιχειρήν, ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εκεί ακριβώς πιστεύω ότι πρέπει να στοχοθετήσουμε τα συστήματά μας ώστε να προαχθεί η ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία. Μόνο ανταγωνιστικές και καινοτόμες επιχειρήσεις μπορούν να ανταγωνιστούν σε παγκοσμιοποιημένες αγορές και μπορούν να επιτύχουν την ανταγωνιστικότητα, τον ανταγωνισμό με επιτυχή τρόπο για να καλύψουν τις ανάγκες των καταναλωτών στις εθνικές αγορές. Θα πρέπει να δούμε αν θα υπάρξουν κάποια κίνητρα ή ελαφρύνσεις φορολογικές ή κάποιες άλλες ε, ευκαιρίες. Όταν βέβαια έρχεται η ώρα δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, φυσικά πρέπει να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης, αλλά σε τοπικό επίπεδο. Δημιουργούνται θέσει απασχόληση σε μια οικονομία. Όσο πιο ανταγωνιστική είναι μια οικονομία λοιπόν, τόσο μεγαλύτερο το επίπεδο, αυξημένο το επίπεδο σταθερότητα. Και εν συμπεράσματι, πρέπει να ξαναγυρίσουμε στι ρίζε τη ευρωπαϊκή κοινότητα στις ρίζες μας και θα πρέπει να αντιληφθούμε, να κατανοήσουμε γιατί δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα τότε στο παρελθόν. Πρέπει να ενδυναμώσουμε τις ε, δικές μας ε, δυνατότητες επαφών ε, για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ και τώρα θα λάβει τον λόγο ο κύριος από το, την Βουλή των Ελλήνων. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κρίση την οποία ζει ο πλανήτης μας είναι πρωτόγνωρη είναι περισσότερο διαρθρωτική, λιγότερο κυκλική και αποτελεί φαινόμενο πρωτοφανές. Βεβαίως όλοι γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει τίποτε κακό χωρίς μέσα του να περιλαμβάνει και κάτι το καλό. Χωρίς να θέλω να λέω ζήτω η κρίση ή να χειροκροτώ την κρίση όπως όλοι μας, η κρίση όμως αναδεικνύει από μόνη της και μια καλή πλευρά Καλή πλευρά βεβαίως εντός των εισαγωγικών. Αγαπητοί συνάδελφοι, με την κρίση μετράμε, θεωρώ πρώτον το πολιτικό μας ανάστημα να διαχειριστούμε αυτή την ίδια την κρίση. Δεύτερο, μετράμε το οικονομικό μας βάθος και εύρος σε σχέση με τα εφιστάμενα μείγματα οικονομικής πολιτικής των χωρών αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταυτόχρονα. Επίσης βλέπουμε τις πραγματικές μας δυνάμεις ως οικονομίες, ως επιχειρήσεις και πάει λέγοντας. Ακόμα η κρίση μας οδηγεί να δείξουμε πραγματικά πόσο ευαίσθητοι είμαστε, πόσο η Ευρώπη και οι χώρες κράτη-μέλη έχουν κοινωνικό πρόσωπο και ακόμη προκαλεί ενδιαφέρον όλο του πλανήτη να δούμε πόσο μεγάλη αντοχή έχει αυτό που όλοι λένε και υποστηρίζουν ως το σωστό ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Αγαπητοί συνάδελφοι, μια φράση κατά μια λογική και κατά κάποια έννοια θεωρώ ότι η κρίση έβαλε τα πράγματα στη θέση τους στην πραγματική τους διάσταση. Βλέπω λοιπόν ότι είναι αναγκαίο και με αυτό θα κλείσω ότι στη σημερινή μας ε, συζήτηση και λογική θα πρέπει να πάμε κόντρα σε αυτό που η, η ίδια η κρίση συχαίνεται και είναι ο αυτοσχεδιασμός. Πρέπει να πάμε προς τον συντονισμό, τη συνεννόηση, μακριά από την πρόσκαιρη γοητεία του προστατευτισμού, να βρούμε τη σωστή δοσολογία για τα κίνητρα, να σταθούμε με διαφάνεια, ξεριζώνοντας τις τάσεις του χρηματοπιστωτικού συστήματος, το οποίο ζητά αύξηση κινδύνων και όχι μόνο. Με μια φράση τελειώνω, χρειαζόμαστε σχέδιο και ιδιαίτερη σοβαρότητα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Και είναι σημαντικό τώρα ο κύριος Λάρσον από το Πανεπιστήμιο Λούντ. Παρακαλώ, για να σχολιάσει τις παρεμβάσεις. Um, Ευχαριστώ. Κάποιες ε, σύντομες παρατηρήσεις. Συμφωνώ εμπολής με αυτά που ελέγχθησαν για τα βασικά μηνύματα αν θέλετε που πρέπει να περάσουν για τη φύση της κρίσης, για την ανάγκη να δρα... αναλάβουμε δράση για τη σημασία που έχει ο συντονισμός των μέτρων του ώστε να αποφευθεί ο προστατευτισμός για την ανάγκη επένδυσης στην έρευνα γιατί πρόκειται για μακροπρόθεσμους στόχους εδώ και τα λοιπά. Θα ήθελα να σχολιάσω αυτό που είπε ο κ. Χάρμπορ για τις ε, ε, άμεσες ε, ε, επεμβάσεις που χρειάζονται. Σήμερα το πρωί διάβασα ότι η Eurobusiness προτείνει ένα πακέτο μέτρων της τάξης του 3,5% του ΑΕΠ όταν οι επιχειρήσεις ζητούν τέτοιου μεγέθους ενέσεις. Αυτό είναι ένα σημάδι ότι πρέπει να δράσουμε, να ανασκουμποθούμε και να υπολογίσουμε ενδεχομένως αν δεν κάνουμε τίποτε τι θα, ποιο θα είναι το κόστος και αν κάνουμε κάτι ποιο είναι το κόστος πάλι. Υπάρχουν αυτά τα πακέτα μέτρων για υποκίνηση και υποδάβληση αν θέλετε της οικονομίας αλλά βλέπουμε ότι τα πακέτα αυτά δεν δουλεύουν, δεν λειτουργούν σωστά. Θα πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη μας. Ε, ψάχνουμε στο σκοτάδι όλοι μας κανείς δεν έχει πείρα κανείς δεν έχει ξαναζήσει μια τέτοια κρίση είναι πρωτόγνωρη η κρίση και το νέο κεφάλαιο του, στο καινούριο βιβλίο του Greenspan το οποίο εκδόθηκε πέρσι λέει, ότι η, η ότι ξεπεράστηκαν τα πιο δύσκολα. Αυτό έλεγε ο Άλαν Γκρίνσπαν πέρυσι το καλοκαίρι. Ε, σας αφήνω να σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι σαν την τωρινή κρίση. Τώρα για τη μαύρη τρύπα, όντως ε, εάν δεν αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της μαύρης τρύπας σωστά δεν έχουμε ελπίδες αλλά και εδώ δεν υπάρχει ε, πείρα σχετική για τα ε, από την ε, αρχές δεκαετίας του 90 έχουμε ε, όμως για τα τοξικά προϊόντα ε, τα τοξικά τραπεζικά προϊόντα ε, και τότε βεβαίως εθνικοποιήθηκαν, κρατικοποιήθηκαν οι τράπεζες και το πρόβλημα η λύση. Αλλά με ιδιωτικές τράπεζες είναι πάρα πολύ δύσκολο να ε, γίνει αυτό. Και ε, πώς είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των τοξικών προϊόντων όταν να δίνουμε βοήθεια σε αυτούς, στους managers οι οποίοι ουσιαστικά απέτυχαν στο έργο τους στις τράπεζες. Όπως είπε ο κάνει ε, πρέπει κάτι να κάνουμε αλλά δεν ξέρουμε τι να κάνουμε και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι μιλάμε για τη χειρότερη κρίση που έχουμε δει στο, τα χρόνια που ζούμε Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστούμε όλοι κύριε Λάσεν για αυτή την ε, εμπεριλήψη συμπερασματική τοποθέτηση και τώρα θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Πιέρ Λεκίγε από την ε, Γαλλική Εθνοσυνέλευση να μας προσφωνήσει. Για πέντε λεπτά διακόπτουμε τη συζήτηση. Θα μας προσφωνήσει επί πεντά λεπτό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρώπη, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά σήμερα, θα πρέπει να αντιμετωπίσει μία μακρά περίοδο οικονομικής δραστηριότητας ε, ε, που θα είναι επιβραδυμένη. Βέβαια όμως μπροστά σε αυτή την, την κρίση οι Ευρωπαίοι πολιτικοί και οι υπεύθυνοι έδειξαν ότι μπορούν να λειτουργήσουν μαζί, ε, να συνεργαστούν αποτελεσματικά. Αυτή είναι μια πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουν όμως όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Κατά τη ε, διάρκεια της Γαλλικής Προεδρίας φάνηκε ποια είναι η προστιθέμενη αξία της Ευρώπης. Το δεύτερο εξάμεινο του 2008 η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μπόρεσε να συντονίσει αποτελεσματικά τα μέτρα υποστήριξης ε, του οικονομικού τομέα. Η συνάντηση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών, ε, η έκτακτη συνάντηση του Ευρωγκρούπ, η Σύνοδος Κορυφής που οργάνωσε η Γαλλική Προεδρία κατάφεραν να κάνουν μια διάγνωση και μια θεραπεία συντονισμένη αν θέλετε. Βέβαια όμως όπως και οι άλλες χώρες και η Γαλλία υπέβαλε το εθνικό της πρόγραμμα ε, για την ε, ενίσχυση των τραπεζών ε, και των προβληματικών τομέων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρώντας ότι θα έπρεπε να σέβεται προφανώς και τους κανόνες, τους ευρωπαϊκούς κανόνες. και ακόμα συζητείται το θέμα από την γαλλική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να επιμείνω σε αυτό, διότι όπως είπε και ο συνάδελφος Σέος Πουανιό, ακούστηκαν διάφορες παρατηρήσεις, ε, κυρίως από τον φίλο μου από την Πολωνική ε, Βουλή. Δεν ε, θεωρώ ότι δεν είναι δίκαιο να κατηγορούμε τα πρόσφατα μέτρα που εξήγηλε η Γαλλία ως προστατευτικά. Θα ολοκληρωθούν και θα εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα όταν και εφόσον ολοκληρωθεί ο διάλογος με την Ευρωπαϊκή αυτό θέλω να το τονίσω γιατί υπήρξαν διάφορες καρικατούρες, διάφορα αστεία. Ποτέ ο Γάλλος πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν ζήτησε να επιστρέψουν τα εργοστάσια ε, αυτοκίνητο, της αυτοκινητοβιομηχανίας ε, που βρίσκονται εκτός Γαλλίας στη Γαλλία. Ποτέ ε, δεν ε, ζήτησε ο Γάλλος πρόεδρος ε, να ε, εφαρμοστούν προστατευτικά μέτρα. Σύμφωνα με το Συμβούλιο της προηγούμενη, του προηγούμενου Δεκεμβρίου χρειαζόμαστε έξυπνα μέτρα τα οποία θα είναι προς όφελος όλων των ευρωπαϊκών χώρων. Να διευκολύνουμε την, την αγορά νέων αεροπλάνων από όλες τις αεροπορικές εταιρείες, αεροπλάνα που θα είναι πιο αποτελεσματικά στον ενεργειακό τομέα, να επενδύσουμε στα καθαρά αυτοκίνητα, να αυξήσουμε την ε, δημιουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ε, να διευκολυνθεί η αγορά κατοικιών, να προετοιμάσουμε την ανταγωνιστικότητα του αύριο με εστιασμένες επενδύσεις ε, που θα προγραμματιστούν για μια διετία το, το πρόγραμμα το οποίο προτάθηκε το Νοέμβριο και υιοθετήθηκε το Δεκέμβριο από τα κράτη-μέλη αποτελούν το πρώτο στάδιο των συντονισμένων εθνικών μέτρων και τα επόμενα ε, συμβούλια της Ευρώπης, ε, θα, τα επόμενα συμβούλια, ευρωπαϊκά συμβούλια θα πρέπει να τα ε, εφαρμόσουν και να τα προωθήσουν. Ε, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια σοβαρή πρόκληση που είναι η εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη στο γεγονός ότι όλες οι συντονισμένες μας δράσεις σε όλα τα κράτη-μέλη αλλά και που ελήφθησαν συντονισμένα και από τους 27 και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι προς όφελος όλης της Ευρώπης. Η εμπιστοσύνη των εταίρων μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι αναδυόμενες χώρες, η ΙΠΑ, η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ρωσία, χώρες προς τις οποίες, τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση στο επόμενο G20 και ε, εκεί θα πρέπει να κάνει και έναν, έναν απολογισμό των ενεργειών μας. Εκεί θα πρέπει να ε, επανατοποθετηθεί ο καπιταλισμός και η θέση μας σε μια διεθνή ανταγωνιστική αγορά. Διότι η Ευρώπη έχει υποχρέωση να επηρεάσει την, τις λύσεις που θα υιοθετηθούν για τα προβλήματα αυτά και ε, θα πρέπει οι λύσεις αυτές να ξεπερνούν τα σύνορά της. Εγώ χαίρομαι για την ταχύτητα με την οποία αντιμετώπισε η Ευρώπη την πρόσφατη κρίση. Στην, στη σύνοδο που έχουν εξαγγείλει, που, που έχει εξαγγείλει η Τσεχική Προεδρία θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλα τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν θα είναι συντονισμένα και όχι προστατευτικά. Θα πρέπει να υπάρξει μια ενιαία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην, στο Λονδίνο στην συνάντηση των G20 γιατί πρέπει για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση η οποία είναι αντάξια της κρίσης του 1929 και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και την σταθερότητα του ευρώ που ε, μας, μας επέτρεψε να μην αντιμετωπίσουμε το διεθνές οικονομικό κράχ του 1929. Πρέπει όμως να είμαστε, να είμαστε σε επιφυλακή. Γιατί, όπως είπε ο κύριος Λάρσεν, η κρίση αυτή είναι σοβαρότατη και λαμβάνοντας υπόψη την ανεργία που ανεβαίνει στη ΣΥΠΑ, στις Ηνωμένες, στην, ε, στην Ιαπωνία και στην Ευρώπη ακόμα, λαμβάνοντας υπόψη την επιβράδυνση της οικονομίας στην Κίνα κυρίως το εύρο ε, της ε, ευρωπαϊκής αντιμετώπισης, η ταχύτητα επιβάλλονται. Και θα ήθελα να επαναλάβω τα λόγια του Ρούσβελτ. Ένα πράγμα μόνο πρέπει να φοβόμαστε. Τον ίδιο το φόβο. Επομένως, ας συνεργαστούμε, ας δουλέψουμε χέρι με χέρι και ας δείξουμε εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον και να συγχαρώ τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Πέπερινγκ, αλλά και την Τσεχική Προεδρία, διότι οργάνωσαν αυτή τη συζήτηση ανάμεσα στα Εθνικά Κοινοβούλια και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι αν υπήρχε ένα θέμα το οποίο έπρεπε να συζητήσουμε μαζί, γιατί αφορά και τις εθνικές πολιτικές αλλά και την Ευρώπη και το συντονισμό των ευρωπαϊκών πολιτικών έπρεπε να το συζητήσουμε μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα λάβει τώρα τον λόγο το μέλος ε, της Βουλής της Σουηδίας, ε, παρακαλώ. Έρενσον. Σα Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση να μπορέσω να συμμετάσχω σε αυτή την κοινή κοινοβουλευτική συνάντηση και να δώσω μια σύντομη τοποθέτηση δήλωση για το σχέδιο ανάκαμψης από πλευρά της Σουηδίας. Ο Σουηδικός Προπολογισμό του 2009 είχε εισαγάγει έναν αριθμό μεταρρυθμίσεων και προγραμμάτων για να απαμβληθεί η οικονομική συρρήκνωση όπως ε, και ε, ε, κίνητρα όσον αφορά τη φορολογία, μείωση φορολογίας όσον αφορά και τις κοινωνικές εισφορές από πλευράς των εισφορών εργαζομένων. Επίσης και στον τομέα των υποδομών, επικέντρωση στον τομέα της παιδείας, κατάτησης έρευνας, προώθηση κοινωνικών μεταρρυθμίσεων και δράση στον τομέα του περιβάλλοντος για τις κλιματικές αλλαγές. Διάφορα από αυτά τα μέτρα θα αντισταθμίσουν σίγουρα, αναμένουμε, την οικονομική αυτή κρίση και η ανάγκη για να υπάρξει ε, καλύτερη απασχόληση, ιδιαίτερα όσον αφορά και την κατάτηση και παιδεία για την απασχόληση και την έρευνα, καθώς επίσης και προοπτικές για την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία οικονομική μακροπρόθεσμα. Τώρα, οι μεταρρυθμίσεις ε, που προβλέπονται από τον προϋπολογισμό και τα μέτρα τα οποία υιοθετούνται για τα επόμενα χρόνια είναι από τα εκτενέστερα μέτρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνολικά, από κοινού με τα μέτρα που ελήφθησαν το 2008 το φθινόπωρο και από κοινού με τον Ιανουάριο εφέτος, έχουμε πάνω από 4 δις ευρώ. Και αυτό αντανακλά περίπου 1,4% του ΑΕΠ της Σουηδίας. Η Σουηδία κατά την τελευταία δεκαετία είχε ε, υγιή δημοσιονομικά θεμέλια με πλεόνασμα και μείωση του ε, χρέους. Με την οικονομική αυτή κρίση όμως ε, τα δημοσιονομικά μας θα επιδεινωθούν τα επόμενα χρόνια και τα δημοσιονομικά ελλείμματα περίπου 1% του ΑΕΠ αναμένονται το 2009 σε αυτό το επίπεδο και το 2010. Η συνολική λοιπόν εκτίμηση, αποτίμηση είναι ότι αυτά τα ελλείμματα είναι προσωρινά και μπορούν να ελεγχθούν. Όμως για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της χρηματοοικονομικής κρίσης, ήδη το φθινόπωρο του 2008 η Σουηδική κυβέρνηση έδωσε προτεραιότητα σε άμεση γοργή δράση για να μπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά οι χρηματοοικονομικές αγορές, ιδιαίτερα η πιστοτική αγορά για την διάθεση δανείων και πιστώσεων. Όπως και οι άλλες τράπεζες, η Riksbank, η Σουηδική Κρατική Τράπεζα από το Σεπτέμβριο 2008 από το 4,75% κατέληξε σε 1% όσον αφορά τα επιτόκια και είχαμε μείωση περαιτέρω όσον αφορά τα επιτόκια που προβλέπεται να σημειωθεί εφέτος. Και όσον αφορά την ε, ζήτηση, όσον αφορά και την διάθεση ρευστότητας, η Riksbank και το ε, Εθνικό Γραφείο για το Χρέο ε, έχουν προβλέψει την διάθεση κυβερνητικών ομολόγων και την δυνατότητα να υπάρξει επένδυση σε αυτές τις δράσεις ήδη από το φθινόπωρο του 2008. Για να υπάρξει ασφάλεια των επενδυτών αυξήθηκαν οι εγγυήσεις ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λάβαμε λοιπόν αυτά τα μέτρα για να διαθέσουμε τώρα, να προβλέψουμε την σταθερότητα και να υπάρξει εμπιστοσύνη στις χρηματοοικονομικές αγορές. Ένας νέος νόμος εγκρίθηκε που θα δίνει την δυνατότητα στην κυβέρνηση να δίνει υποστήριξη για δημοσιονομικές εγγυήσει ε, στα θεσμικά όργανα και με άμεση ε, δραστηριοποίηση. Με αυτό το νόμο ε, υπεγράφει ένα πρόγραμμα εγγυήσεων και ένα ειδικό ταμείο εγγυήσεων δημιουργήθηκε για την λήψη αυτών των υποστηρικτικών μέτρων. Η Σουηδική κυβέρνηση πρόσφατα προανήγγειλε νέα μέτρα για τις τράπεζες για να μπορέσουν να εμπλακούν σε αυτά τα προγράμματα και εξετάζει και περαιτέρω μέτρα για την ενίσχυση της σταθερότητας ε, στην χρηματοοικονομική αγορά όταν αυτό θα είναι αναγκαίο για να αντιμετωπίσουμε την στενοπό της ε, διάθεσης πιστώσεων για τις εξαγωγές ε, είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε δυνατότητες ε, για τις εξαγωγές μας από πλευράς πιστώσεων. Επιπλέον δημιουργήθηκε ένα πλαίσιο εγγυήσεων τέτοιων εξαγωγικών πιστώσεων η χρηματοοικονομική ανάπτυξη και η υπηρεσία υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είχε και εκείνη οι δυνατότητες για αυξημένη δανειοδότηση, διάθεση πιστώσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εν τέλει, για να ενισχύσουμε την φερεγγιότητα και την ρευστότητα ε, έγιναν αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο και όσον αφορά την φορολογία, δίνοντας στους εργοδότες ευκαιρίες ε, για να υπάρξει ανακούφιση όσον αφορά την καταβολή εισφορών ε, ή και αναβολή τους για μια περίοδο το, κατά το μέγιστο 12 μηνών. Και για να μπορέσουμε περισσότερο να δώσουμε δυνατότητες ε, να δραστηριοποιηθεί η αυτοκινητοβιομηχανία ιδιαίτερα όσον αφορά την προστασία του κλίματος και της ασφάλειας ε, δημιουργήθηκε μια υπηρεσία που θα παρακολουθήσει και εκ του σύνεγγυ στην έρευνα στην αυτοκινητοβιομηχανία και θα την τονώσει. Η κυβέρνηση επίσης μπορεί να παράσχει δάνεια για την ε, υποστήριξη επιχειρήσεων με αντίστοιχες εγγυήσεις για τις αυτοκινητοβιομηχανίες που αντιμετωπίζουν ε, πιέσεις και δυσκολίες. Και αυτά τα μέτρα φυσικά υιοθετήθηκαν πάντα ε, ευθυγραμμιζόμενοι με το πλαίσιο της, των απαιτήσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη ρύθμιση των θεμάτων επιδοτήσεων από την Ευρωπα... τις Ευρωπαϊκές Αρχές. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας ευχαριστώ. λέει ο πρόεδρος. Θα ήθελα να καλωσορίσω τώρα τον προεδρεύοντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και πρωθυπουργό της Τσεχικής Δημοκρατίας τον κύριο Τοπολάνεκ, Μίρεκ Τοπολάνεκ. Říkali, že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 Ίσως ε, είναι για να έχουμε μεγαλύτερη αγωνία. Thank Dostávám informaci, že v zákulisí pro... Κοιτάξτε, μόλι τώρα μου είπαν ότι υπάρχει ότι γίνεται συζήτηση μεταξύ του Προέδρου του Κοινοβουλίου α, ε, κυρίου Πέτερινγκ, του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του κυρίου Μπαρόζο και του Προέδρου του Συμβουλίου του κυρίου Τουπολάνεκ. Α, ε, Κρίμα, φαντάζομαι ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα, αλλά θα προτιμούσαμε οι τρεις αυτοί κύριοι να ήταν στη δική μας εδώ, εντός αιθούσης.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 βρίσκεται μαζί μα εδώ ο Προεδρεύων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Πρωθυπουργό τη της Δημοκρατία ο κ. Στοπολάνεκ. Χαιρετίζω και τον κύριο Παρόζο, ε, τον Πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Δίνω τον λόγο στον Πρόεδρο τη ε, βουλή της χώρας μου, τον κύριο Βουλτσέκ. και το λόγο στον κύριο Τοπολάνεκ. Κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε του Κοινοβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η σημερινή συνάντηση, διακοινοβουλευτική συνάντηση, σήμερα κατά τύχην γίνεται η συνειδητά γίνεται μερικές μέρες πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων που θα γίνει στις αρχές Μαρτίου. Το θέμα βεβαίως είναι η πιο σοβαρή οικονομική κρίση που έχουμε αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια και μια κρίση για την οποία ξέρουμε ότι δεν είναι μόνο τα κράτη-μέλη που πρέπει να αναζητήσουν τις λύσεις αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις και τα ε, κοινοβούλια των χωρών μελών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλοι βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση και θα πρέπει να αναζητήσουμε λύσεις. Ξέχασα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης των διαφόρων κρατών μελών που βρίσκονται και αυτά στην ίδια ε, κατάσταση. Ε, είμαστε όλοι στο, στην ίδια βάρκα στο κάτω κατάστρωμα, στο πάνω κατάστρωμα, είμαστε στον Τιτανικό, ε, βυθιζόμεθα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι λένε ότι θα πρέπει να προσφύγουμε στον προστατευτισμό υπάρχουν λοιπόν και κάποιοι εθνικιστές οι οποίοι χοροπηδούν από τη χαρά τους ε, στο <coughs> τιτανικό αυτό που βασίζεται ε, είναι γρήπη η κρίση ή είναι επιδημία πανευρωπαϊκή πανδημία για να μην πω επιδημία είναι ε, η κρίση αυτή είναι μια κρίση που μπορούμε να τη δείχνουμε από το δάχτυλό μας να πούμε ότι είναι αυτό το κακό το οποίο δημιουργεί το πρόβλημα την ξέρουμε την κρίση όλα αυτά οδήγησαν στο να συγκαλέσουμε στις αρχές Μαρτίου ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των αρχικών, αρχικών κρατών και κυβερνήσεων ένα έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να συναντιόμαστε πιο συχνά για να μπορούμε να ε, συζητήσουμε περισσότερο τα πράγματα γιατί μας χρειάζονται συχνότερες συζητήσεις και μάλιστα σε ψηλό επίπεδο δεν λέω ότι σε χαμηλότερο επίπεδο, σε υπουργικό επίπεδο ή ακόμη και επίπεδο ομάδων εργασίας δεν γίνεται δουλειά όμως η κρίση την οποία αυτή τη στιγμή διατρέχουμε είναι κρίση εμπιστοσύνης σε μεγάλο βαθμό α, μπορεί να εκφράζεται ποσοτικά με κάποιους αριθμούς αλλά έχει και πάρα πάρα πολύ έντονες πολιτικές διαστάσεις όπως όλες οι σοβαρές κρίσεις το να ξεπεράσουμε λοιπόν την κρίση ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και, αλλά δεν είναι σημαντικό μοναχά για τις επιχειρήσεις είναι σημαντικό και για τις κυβερνήσεις οι οποίες ε, μόνο αν ξεπεράσουν την κρίση θα επιβιώσουν η κρίση θα διαρκέσει πολύ ναι εάν δεν καταφέρουμε να συμφωνήσουμε όλοι μαζί σεβόμενοι τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού και της ε, ε, εσωτερικής ε, ε, αγοράς δεν θα τα καταφέρουμε θα χάσουμε όλοι αν ακολουθήσουμε τους κανόνες του προστατευτισμού και του μαρκαντιλισμού αν πέσουμε σε, αυτή την παγίδα και πιστεύω ότι η πολιτική διάσταση της κρίσης ίσως τελικά ε, αποδειχθεί σοβαρότερη της οικονομικής διάστασης. Και είναι σημαντικό λοιπόν εν ώψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του των αρχών Μαρτίου να έχουν γίνει σχετικές συζητήσεις και να, έχει ακουστεί η να έχουν ακουστεί οι απόψεις όλο και περισσότερων. Ε, όταν εγώ είχα ε, ε θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε λοιπόν ότι θα έχουμε δύο Ευρωπαϊκά Συμβούλια εαρινά φέτος. Ένα στις αρχές Μαρτίου για το θέμα της οικονομικής κρίσης, για τα οικονομικά θέματα και ένα άλλο το Μάιο για την απασχόληση. Η... Το στις 10 Φεβρουαρίου οι Υπουργοί Οικονομικών είπαν ότι πρώτα πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα τοξικά προϊόντα των τραπεζών που δημιουργούν όλο και μεγαλύτερα προβλήματα και δεύτερον να εξασφαλίσουμε ότι θα αρχίσει και πάλι ο τραπεζικός δανεισμός ε, εδώ βεβαίως βλέπουμε την ε, στενή σύνδεση των ε, ε, οικονομικών με τις πολιτικές διαστάσεις. Δεν μπορούμε από τη μια στιγμή στην άλλη να μειώσουμε τα επιτόκια για να αρχίσουν να δανείζουν και πάλι οι τράπεζες. Οι τράπεζες φοβούνται την αστάθεια, φοβούνται την ανασφάλεια και αν δεν αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στο γενικότερο κλίμα οι τράπεζες δεν θα μπορέσουν να αντιδράσουν σωστά. Πρέπει λοιπόν και εμείς οι πολιτικοί να ανασκουμποθούμε εδώ. Από την άλλη μεριά οι επιχειρήσεις ε, οι οποίες καλούνται να παράγουν χωρίς κέρδος γιατί δεν τραβάει η αγορά τα προϊόντα τους ή γιατί ε, ο κόσμος δεν μπορεί να ξοδέψει ε, και αυτές οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε κίνδυνο προφανώς τα οποία πρέπει να ξεπεραστούν και όλες οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουν πρόβλημα όλες οι κυβερνήσεις των χωρών μελών και οι μικρές και οι μεγάλες ωστόσο ο κίνδυνος να πέσουμε στην παγίδα του ε, προστατευτισμού είναι μεγάλος και θα ήθελα σχετικά να σας πω ένα ανέκδοτο από το Σοσιαλιστικό Κόμμα ένας συνάδελφος από μια ομάδα εργασίας είπε στον, σε έναν υπουργό ε, φοβόμαστε ότι όταν μιλάτε για αγορά ε, κύριε Υπουργέ εννοείται ελεύθερη αγορά καταλαβαίνετε τι εννοώ ελπίζω φίλες και φίλοι θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι πρέπει να υπάρχει διεθ... παγκόσμια κατανομή εργασίας. Οι αρχές της κοινότητας πρέπει να τηρούνται. Και ο φόβος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 ότι οι υπηρεσίε αξιολόγηση οι παγκόσμιε θα κρίνουν αν η οικονομία μας, οι οικονομίες μας ε, περισσότερο ότι δεν, είμαστε, δεν βρισκόμαστε στο επίπεδο που βρισκόμαστε μέχρι τώρα έχουμε προβλήματα και σαν κυβερνήσεις πλέον να δανειστούμε όλα αυτά αυτά συμβαίνουν για όλους και γι' αυτό ο μόνος δρόμος μπροστά είναι μαζί. Θέλουμε να υπάρχει δημοσιονομική πειθαρχία, θέλουμε να τηρούνται οι όροι του Συμφώνου Σταθερότητας α, γρήγορα, να, να επανέλθουμε σε μια σταθερότητα γρήγορα στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό και τη στιγμή που αυτό είναι ε, δυνατό η Κομισιόν είναι ο θεματοφύλακας των βασικών ε, των ε, αρχών της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και θέλουμε να κάνει το καθήκον της αλλά πρέπει και εμείς να κάνουμε το καθήκον μας για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τη κρίση γρήγορα να μην πρόκειται για μία υπερβολικά μακροπρόθεσμη ε, μακρά κρίση όπως ήταν η κρίση του 29 θέλουμε να Ε, ε, αγωνιστούμε όλοι μαζί ε, και δεν θα ήθελα να σας δακτυλοδείξω αυτή τη στιγμή εσάς ε, τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά εν και των ευρωπαϊκών εκλογών του Ιουνίου θα ήθελα να πω ότι πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα στις υποσχέσεις που δίνετε διότι αν κάνετε υποσχέσεις που δεν, δεν μπορούν να τηρηθούν ε, υπονομεύεται ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη του κόσμου ελευθερία αλληλεγγύη ε, είναι οι βασικές μας αρχές αυτές θα πρέπει να υποστηρίξουμε ε, και ελπίζω ότι όλοι ενωμένοι θα προχωρήσουμε προς την υποστήριξη αυτών των ευρωπαϊκών αρχών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρωθυπουργέ το Πολάνεκ για τη δική σας παρέμβαση και συνεισφορά στις σημερινές μας διαβουλεύσεις. Τώρα θα δώσω τον λόγο στον Πρόεδρο Μπαρόζο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Πρωθυπουργέ, Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κύριε Μιρέκ, κυρίες και κύριοι βουλευτές η χρηματοπιστωτική κρίση και η οικονομική κρίση που πλήττει την Ευρώπη σήμερα μας αναγκάζει να συντονίσουμε όλες τις πολιτικές και όλες τις ενέργειες των θεσμικών παραγόντων, των κοινωνικών εταίρων, των ε, κυβερνήσεων. Για αυτούς τους λόγους ακριβώς το να κινητοποιήσουμε και να συντονίσουμε δηλαδή ε, μας ανα, ε, αναγκαστήκαμε να ξεκινήσουμε μια σειρά συναντήσεων πάρα πολύ σημαντικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη-μέλη και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θα πρέπει να εξετάσουν περάσουν από κοινού όλα τα μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα για να αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι μια βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποκλείονται βέβαια η εθνικοί οι εθνικισμοί, οι οικονομικοί εθνικισμοί και οι προστατευτισμοί. Διότι είδαμε αυτά τα μέτρα πόσο επιδεινώνουν την κρίση. Θα πρέπει να συντονίσουμε τα, ε, τα μέτρα ανάκαμψης έτσι ώστε να μην υπάρχουν δεσμενείς επιπτώσεις για τα άλλα κράτη. Αυτή είναι μία από τις βασικές αρχές της ενιαίας αγοράς. Το Συμβούλιο ε, το Ευρωπαϊκό στις 19 ε, Μαρτίου θα είναι ένα σημαντικό βήμα, διότι θα, μετά την άτυπη συνάντηση κορυφή τη 1η Μαρτίου ε, θα ε, ξεκινήσουμε μια νέα πορεία και θα, η οποία θα ολοκληρωθεί επίση και με τη συνάντηση του Μαΐου που θα αφορά την απασχόληση. Επίση ε, θα πρέπει να συντονίσουμε και την στάση μα εν ώψη τη συνάντηση στο Λονδίνο στι 2 Απριλίου. Αυτό θα το κάνουμε και στο Βερολίνο μετά από πρόσκληση τη καγκελαρίου κυρία Μέρκελ. Θα πρέπει επομένως να ξεκινήσει μια νέα εφαρμογή και επιβολή κανόνων και είναι προφανές ότι σε αυτή την πορεία θα πρέπει να συμμετέχουν και οι εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων. Θα προσπαθήσουμε να τελειοποιήσουμε το, το σύστημα ανάκαμψης το οποίο ξεκίνησε η Κομισιόν τον Νοέμβριο και χαίρομαι ιδιαίτερα μπορώ να συζητάω σήμερα μαζί σας. Κυρίες και κύριοι, αντιμετωπίσαμε άμεσα στην κρίση. Οι παρεμβάσει ε, των ε, κυβερνήσεων το φθινόπωρο του 2008 μας έκαναν να αποφύγουμε, μας επέτρεψαν να αποφύγουμε την ε, κατάρρευση και ε, ήταν αποτελεσματικά τα μέτρα αυτά, διότι ελήφθησαν συντονισμένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπό την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να, έχουν, να υπάρχει πίστοση, αν θέλετε, στις επιχειρήσεις ε, με, ε, με κανονικά επιτόκια. Και θα πρέπει να δούμε πόσο αντιμετωπίζουμε τα, προ, τα προβλήματα των τραπεζών. Και η, θα χρειάζεται ευρωπαϊκή προσέγγιση, η οποία θα καθοδηγήσει τις εθνικές πολιτικές Επίσης ε, θα πρέπει να εξετάσουμε και να σχεδιάσουμε τον, το μέλλον του χρηματοπιστωτικού τομέα. Με μία βασική αρχή. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές ε, θα πρέπει να ε, ανακαλύψουν την αρχική τους, τον αρχικό τους στόχο που ήταν να εξυπηρετήσουν την οικονομία όλων. Θα πρέπει να υποστηρίξουν μια βιώσιμη και αποτελεσματική οικονομία. Πώς θα γίνει αυτό όμως η ομάδα Ντελαροζιέρ θα μας υποβάλει μια έκθεση ε, σε λίγο και με βάση την έκθεση αυτή θα υποβάλω προτάσεις στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επειδή οι χρηματοπιστικές αγορές είναι σφαιρικές, είναι παγκόσμιες, ε, θα πρέπει και οι λύσεις μας να είναι ε, παγκόσμιες. Δηλαδή θα πρέπει για τα παγκόσμια προβλήματα να αντιμετωπίσουμε παγκόσμιες, να παγκόσμιες λύσεις. Και κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Προεδρίας ο πρόεδρος Αρκοζή και εγώ πήγαμε στην Αμερική και συναντήσαμε να, και προτείναμε να οργανώσουμε αυτή τη σύνοδο κορυφής όπου εκεί ακούστηκε η φωνή της Ευρώπης. Γιατί, Γιατί είμαστε ενωμένοι όλα τα 27 κράτη-μέλη αποφάσισαν να υιοθετηθεί μια συνακτική θέση εκ των προτέρων και είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσουμε και άλλη μια φορά μια ε, συντονισμένη θέση και για τη συνάντηση την Τεαρινή στο Λονδίνο, τον, τον G20. Η, εμείς υιοθετήσαμε τον Δεκέμβριο του 2008 ένα φιλόδοξο σύστημα ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας, το οποίο προετοίμασε η Κομισιόν και το ενέκριναν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Φορολογικά κίνητρα δόθησαν για την ε, περίοδο μέχρι το 2010. Ε, θα είναι 3,3% του ΑΕΠ ΑΕΠ και θα φτάσει για να μην πω και 4% του ΑΕΠ. Αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια. Ιστορικά είναι εκπληκτική προσπάθεια την οποία να καταβάλουμε αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι ήταν και η σωστή κίνηση διότι ο ιδιωτικός τομέας είναι αδύναμος. Επομένως το δημόσιο πρέπει να καλύψει το κενό και ήταν, είναι λογικό να συντονίσουμε αυτή την, ε, ε, δημόσια, τις δημόσιες κινήσεις αν θέλετε σε ευρωπαϊκό επίπεδο χρειάζεται συντονισμός γιατί με τον τρόπο αυτό τα κράτη-μέλη θα μπορούν να υποφεληθούν και από τα μεμονωμένα τα εθνικά προγράμματα ανάκαμψης της οικονομίας διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κατάσταση στις 27 χώρες είναι διαφορετική. Από την άλλη πλευρά δεν είναι μια επιταγή εν λευκό αυτό το, αυτή η πολιτική και αυτά τα φορολογικά κίνητρα τα οποία ε, δίδονται. Θα πρέπει να δούμε ε, ποια είναι τα, πώς θα αντιμετωπίσουμε και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, ποιο, θα είναι, ποιο είναι το hangover θέλετε, του ε, ελλείμματος και θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έτσι ώστε να ε, έχουμε με την, ε, και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και να σταθεροποιήσουμε την ανάπτυξή μας. Και αυτό είναι ένας τρόπος με τον οποίο θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε, να καλύψουμε το χρέος όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Τα κράτη-μέλη πιστεύω ότι κάνουν τις προσπάθειές τους. Έχει ξεκινήσει δηλαδή η εφαρμογή του προγράμματος. Τώρα βέβαια θαύμα από μια μέρα στην άλλη δεν μπορεί να γίνει. Είναι αλήθεια ότι μπορεί βέβαια η κατάσταση να επιδεινωθεί πριν γίνει καλύτερα. Αλλά τέλος πάντων είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι κάποια στιγμή με το πρόγραμμα αυτό ανορθώνοντας την εμπιστοσύνη θα λειτουργήσει το πρόγραμμα, θα ε, ε, υπάρξει μεγαλύτερη ζήτηση ή η Κομισιόν καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε η κοινοτική συνεισφορά να ε, λειτουργήσει ο δυνατόν πιο γρήγορα. Συνεργαζόμαστε με τις κυβερνήσεις και με τις τοπικές αυτοδιοικήσεις έτσι ώστε να συντονίσουμε τις ε, δαπάνες. Ε, θέλουμε να έχουμε μια πιο αποτελεσματική παρέμβαση. Επίσης υποβάλαμε προτάσεις έτσι ώστε τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία δεν είχαν χρησιμοποιηθεί από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό να προσανατολιστούν προς τον ενεργειακό τομέα. Είμαι σίγουρος ότι θα καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία διότι είναι εστιασμένες οι επενδύσεις αυτές. Με τον τρόπο αυτό με ένα σμάρο δύο τριγώνια. Όχι μόνο θα ενισχύσουμε την οικονομία, αλλά θα αυξήσουμε και την ενεργειακή μας ασφάλεια, που είναι ε, μια βασική προτεραιότητα, ε, λαμβάνοντας υπόψη και την, ε, τα τελευταία προβλήματα που αντιμετωπίσαμε με το φυσικό αέριο. Όμως η βασική μας προτεραιότητα πρέπει να είναι να προστατεύσουμε τους πολίτες μας από την κρίση. Γι' αυτό θα οργανώσουμε τον, τον Μάιο ένα, μια σύνοδο κορυφή για την απασχόληση και χαίρομαι γιατί δέχτηκε την πρότασή μου ο κύριος Στοπολάνεκ να οργανώσει μια σύνοδο η οποία θα είναι εστιασμένη στα προβλήματα ανεργίας και απασχόλησης. Και ελπίζω ότι η σύνοδος αυτή θα έχει αυτά αποτελέσματα. Και ε, θα πρέπει η συζήτηση να εστιαστεί σε τρία θέματα. Η πρώτη προτεραιότητα είναι να διατηρηθούν οι άνθρωποι στις θέσεις απασχόλησής τους, όπου είναι δυνατόν. Υπάρχουν ε, ε, παραδείγματα επιτυχή, όπου βλέπουμε ότι έχουμε βραχυπρόθεσμη επιδότηση για τις θέσεις απασχόλησης και την απόκτηση προσόντων. Αυτό θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να το επαναλάβουμε και να το ενθαρρύνουμε. Διότι θα ήταν ε, λάθο να επιτρέψουμε σε άτομα να χάσουν τη θέση απασχόληση του, απασχόλησής τους γνωρίζοντας ότι κάποια στιγμή αυτές οι εταιρείες θα μπορέσουν να τους επαναπροσλάβουν από τη στιγμή που επιληθεί η κρίση. Αυτό είναι κάτι το οποίο λειτουργεί σε κάποια κράτη-μέλη και είχαμε κάποια καλά αποτελέσματα μέχρι τώρα. Δεύτερον, εκεί που κάποιος χάνει τη δουλειά του, διότι δυστυχώς ε, και αυτό συμβαίνει θα πρέπει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας όσο το πιο γρήγορα τα άτομα αυτά και το πρόγραμμα ανάκαμψής ε, επιτρέπει στα κράτη-μέλη να προσανατολίσουν την, τους πόρους του κοινωνικού ταμείου ή στην ενίσχυση της αγοράς και να προσαρμοστούν να ε, προσανατολιστούν συγγνώμη, τα χρήματα αυτά στα άτομα τα οποία βρίσκονται σε πιο αδύναμη θέση. Τρίτον, οι νέοι τα άτομα αυτά τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολία στα να, να μπουν στην αγορά εργασίας. Εάν η δυσκολία εισόδου στην αγορά εργασίας γίνει μακροπρόθεσμη ενεργεία έχουμε χάσει το παιχνίδι. Πρέπει να βρούμε πολιτικές που θα μας αποτρέψουν, θα αποτρέψουν κάτι τέτοιο. Μην κάνουμε το λάθος για να έχουμε μια βιώσιμη ανάκαμψη θα πρέπει η, αυτά τα μέτρα τα οικονομικά τα οποία δίδονται τώρα, ε, το, η οικονομική ενίσχυση να ε, μετατραπούν σε μια μακροπρόθεσμη πολιτική. Και εδώ μπαίνει και στο παιχνίδι η στρατηγική της Λισαβόνας για την, για την, ε, για την απασχόληση οι, τα διαδροτικά με ταμεία μπορούν να υποστηρίξουν την απασχόληση ε, ε βραχυπρόθεσμα και μπορούν ταυτόχρονα όμως να ε, λειτουργήσουν και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Βέβαια θα πρέπει να είναι τα σωστά μέτρα διότι η εσωτερική ε, αγορά θα πρέπει, η εσωτερική ενιαία αγορά θα πρέπει να παραμείνει ένας βασικός προσανατολισμός για μας. Ο στόχος μας αυτός είναι. Η ιστορία έδειξε ότι ο η εθνικιστική οικονομία και ο προστατευτισμός δεν αποδίδουν. Θα πρέπει επομένως να ε, ε, ε, κλείσουμε τα αυτιά μας και να μην ακούμε τις σιρήνες του προστατευτισμού. Τι κάνει τόσο σημαντικό το ευρωπαϊκό παράδειγμα. Είναι ο σεβασμός του κράτους δικαίου. Και όλοι δεσμευόμαστε από τον νόμο. Το να σεβόμαστε τον νόμο είναι βασική προϋπόθεση για την εξωτερική μας αξιοπιστία. Πώς μπορούμε να προτείνουμε νέους κανόνες για τις παγκόσμιες αγορές. Πώς μπορούμε να ασκήσουμε κριτική σε κάποιους εταίρους μας διότι δεν συμφωνούν με κάποιες βασικές παγκόσμιες αρχές και ταυτόχρονα να μην μπορούμε εμείς να σεβαστούμε τους δικούς μας κανόνες στην εσωτερική αγορά. Εάν το προτείνουμε αυτό για τους υπολείπους, το προτείνουμε διότι η ευρωπαϊκή εμπειρία απέδειξε ότι η αγορά λειτουργεί μόνο εάν υπάρχουν σαφείς κανόνες. Κυρίες και κύριοι, αυτή η κοινή, αυτή, αυτή η συνάντηση ε, ε, κοινοβουλίων είναι ένα σημαντικό θέμα στην ε, ημερήσια διάταξή μου. Και ε, είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι οι συναντήσεις αυτές έχουν κάποια προστιθέμενη αξία. Όπως είπα, έχω πει πάρα πολλές φορές, ε, είτε θα σκεφτούμε μαζί είτε θα βυθιστούμε μαζί. Και νομίζω ότι μπορούμε να κολυμπήσουμε από κοινού και εάν αποφύγουμε οποιαδήποτε προστατευτισμό θα τα καταφέρουμε να βγούμε από την κρίση και να βγούμε και πιο δυνατοί από την κρίση από ό,τι είμαστε πριν. Διότι αυτό περιμένουν οι πολίτες από εμά, ας μην τους απογοητεύσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μπαρόζο για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβασή σας. Θα ήθελα τώρα να ανοίξουμε το δεύτερο μέρος, το δεύτερο γύρο της συζήτησης. Μας παρακολουθούν και από πλευράς της Προεδρίας του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Τέμεσερ τώρα θα λάβει τον λόγο από την Αυστριακή Βουλή. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, όταν παρακολουθεί κανείς αυτές τις παρεμβάσεις ε, χθε το απόγευμα και τις σημερινές σήμερα το πρωί, καταλαβαίνει ότι βρίσκεται κάπου όπου συζητείται πώς μια επικείμενη σύνοδος κορυφής, οικονομική σύνοδος κορυφής ή μια οικονομική κρίση θα μπορούσε να ξεπεραστεί. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε μέσα όμως σε αυτή την κρίση. Δεν είναι επικείμενη. Δεν περνάει ούτε μια μέρα στη εβδομάδα στην Ευρώπη που να μην ε, χάνονται θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη και χιλιάδες κιόλα. Και εμείς συζητούμε εδώ μια μισή ολόκληρη μέρα για το τι θα μπορούσαμε λέει να κάνουμε, τι θα έπρεπε να κάνουμε, τι είναι η ηθική επιταγή να κάνουμε. Κυρίες και κύριοι, δεν τα κάνουμε όμως αυτά. Και γιατί δεν τα κάνουμε. Ξέρετε, ο Μπαράκ Ομπάμα ε, συχνά αναφέρθηκε. Ο Μπαράκ Ομπάμα ούτε ένα μήνα δεν είναι καν στην εξουσία και έχει ένα πακέτο συγκυρία το οποίο ξεκίνησε με 5,5% του Αμερικανικού ΑΕΠ. 780 δις δολάρια και δεν λαμβάνεται καν υπόψη και η αυτοκινητοβιομηχανία που υπό τον Μπούς είχε τεράστιες ε, ε, επιδοτήσεις. Και έτσι μετά από ένα μήνα, ούτε καν ένα μήνα, έχει τεθεί σε ισχύ κιόλα αυτό το πακέτο. Εμεί συζητάμε ακόμα όμω με κάθε σοβαρότητα τι θα έπρεπε να κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν τα κάνουμε όμω. Αν ένα μικρομεσαίο έχει ένα πρόβλημα, υπάρχει σαφή αρμοδιότητα ποιο θα κάνει τι και υπάρχει και χρονοδιάγραμμα για τη δράση. Εγώ θα ανέμενα κατά το τέλο αυτή τη ε, συνδιάσκεψη ε, που με τρει μήνε καθυστέρηση ε, ολοκληρώνεται, θα ήθελα να πω ότι αναμένω από εσά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει το καλό παράδειγμα ω προπομπό, ω πρωτοπόρο. Ο κύριο είπε χθε 1,7% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να διατεθεί για οικονομικά μέτρα. Δηλαδή μεταξύ 200 ή 300 δις ευρώ. Ε, κάντε το αυτό. Στο πρώτο τρίμηνο κιόλας του 2009. Και αν πιστεύετε κύριε Μπαρόζο ότι με μια σύνοδο κορυφής για την απασχόληση μπορείτε να περιμένετε ως τον Μάιο, ε τότε τον Μάιο θα είχε εκατοντάδες χιλιάδες πρόσθετους ανέργους η Ευρώπη. Σας το διαβεβαιώνω αυτό. Και το αν αυτό θα είναι φθηνότερο το αμφισβητώ, το διαμφισβητώ έντονα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενος αγορητής ε, η Βίνσκι από την Πολωνική Βουλή. Σας ευχαριστώ πολύ. Και Κύριε Συμπρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εχθές ο κύριος Τρισέ ανέφερε τρεις πτυχές της κρίσης και τους κύριους λόγους ε, για αυτή την κατάσταση. Η κατάσταση όμως είναι πιο επιδεινωμένη, πιο... είναι χειρότερη από αυτή που νομίζαμε και σύμφωνα με τα περισσινά στατιστικά στοιχεία και τις ε, εκτιμήσεις ε, του βραβευθέντος με το βραβείο Νομπέλ Οικονομίας ε, είναι η δεύτερη βαθιά ύφεση. Πολύ δύσκολο να την ξεπεράσουμε. Είναι μια κρίση του καπιταλιστικού συστήματος. Η πρώτη από την δεκαετία του 1930 κατά τον 20ο αιώνα. Η δεύτερη. Δεν είναι όπως όσον αφορά την Άπο Ανατολή πριν από 10 χρόνια. Είναι μια κρίση του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού αυτή τώρα. Και αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι δεν θα έπρεπε να χάσουμε πια άλλο χρόνο προσπαθώντας να συναγάγουμε συμπεράσματα και να μάθουμε τα σωστά μαθήματα. Πρέπει να δράσουμε άμεσα. Χρειάζεται μια νέα διεθνή τάξη πραγμάτων από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την Ευρώπη συνολικά, αλλά πραγματικά χρειαζόμαστε μια νέα τάξη πραγμάτων για τους 7 δισεκατομμύρια κατοίκους αυτής της οικουμένης, αυτού του ε, κόσμου. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι υπάρχει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Ο πρόεδρος Μπαρόζο ανέφερε τη λέσχη των 20, την G20. Αυτό θα μπορούσε να μας πάει πιο κοντά σε αυτό το πρόγραμμα. Δεν υπάρχει ακόμα αυτό. Οι εθνικές αντιδράσεις ε, και η δραστηριοποίηση σε εθνικό επίπεδο διαφέρει πολύ από κράτος σε κράτος. Και δεν είναι το θέμα εδώ των κατοίκων κατηγοριών των επιβατών σε ένα σκάφος ε, όπως ανέφερε ο πρόεδρος το Πολάνε. Κάποιες χώρες, κάποιες χώρες όπως η Γαλλία επικεντρώνουν στην έρευνα, στην τεχνολογία και τις επιστήμες. Και η πολωνική κυβέρνηση επιλέγει τι δημοσιονομική πειθαρχία και περιστολή. Οι Γάλλοι όμω κάνουν το σωστό πράγμα. Θα έπρεπε να διασφαλίσουμε λοιπόν θέσει απασχόληση. Και γι' αυτό όσον αφορά τη σύνοδο κορυφή στην Πράγα, την άτυπη σύνοδο, είναι πολύ σημαντική σίγουρα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο ρόλο τη επίση έχει θεμελιώδη σημασία όσον αφορά τον έλεγχο και την επιτήρηση. Χρειαζόμαστε λοιπόν σαφεί στόχου συνετούς και καλομελετημένους στόχους. Δεν τους έχουμε αυτή τη στιγμή. Πρέπει να ξεπεράσουμε αυτή την αδυναμία μας στην Πράγα, στο Βερολίνο, στι στις Βρυξέλλες. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση. Σας ευχαριστώ και στη συνέχεια θα λάβει τον λόγο Στένμπεργκ από την Σουηδική Βουλή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ θερμά επίσης και τον κύριο Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μπαρόζο που αναφέρθηκε στι κοινωνικέ πτυχέ και τις πτυχές που αφορούν τους ανθρώπους σε σχέση με τη Σύνοδο Κορυφής για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Καμιά φορά έχω την εντύπωση ότι αυτές τις πτυχές τις ξεχνάμε αυτές τις ε, τελευταίες μέρες. Θα ήθελα να πω, έχω μια ερώτηση, κύριε Λάρσον, να προβληματιστούμε, να δούμε αν μήπως μέσα στο πλαίσιο αυτής της κρίσης θα έπρεπε να μπορέσουμε να συζητήσουμε τι μπορεί να γίνει για το ότι άτομα, πολίτες, ε, ε, ε πολλές φορές ε, επομίζονται υπερβολικά χρέη και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πραγματικά ανθρώπινα δεινά και ανθρώπινη δυστυχία. Σας ευχαριστώ πολύ και στη συνέχεια θα λάβει τον λόγο ο κύριος Βίτεμπροντ από την Πολωνική Βουλή παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας ε, τον Πρωθυπουργό κύριο Τοπολάνεκα της ε, Τσεχικής Δημοκρατίας και τον κύριο Μπαρόζο, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ε, παρεμβάσεις τους ε, και σε αυτή τη συζήτηση. Είναι αισιόδοξε αυτέ οι παρατηρήσει. Συμφωνώ όμω περισσότερο με τον Αυστριακό συνάδελφο που λέει ότι χρειαζόμαστε κατεπήγοντα μέτρα, συνετά καλομελετημένα μέτρα. Στην κρίση, έκδηλη κρίση που αντιμετωπίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκόσμια, αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα μεγαλύτερο βαθμό ανοιχτή προσέγγιση, αλληλεγγύη, εμπιστοσύνη, ανοιχτού χαρακτήρα. Δεν θα έπρεπε να κλειστούμε σε ένα οχυρό και να δημιουργήσουμε τύχη γύρω μα. Η κατεύθυνση που θα ακολουθήσουμε έχει σίγουρα θεμελιώδη σημασία και η προσέγγιση μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης και τους συναδέφους από την Γαλλία που παρενέβησαν. Επειδή επετέχθη συμφωνία υπό την Γαλλική Προεδρία για το πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, για την προστασία του περιβάλλοντος. Και τώρα ήρθε η χρονική στιγμή να τα σεβαστούμε και να τα υλοποιήσουμε όλα αυτά. Επίσης καλωσορίζω, είναι καλοδεχούμενα τα λόγια και οι παρατηρήσει του κυρίου Λάρσον. Προσέξτε, η υλοποίηση, εφαρμογή της στρατηγικής για την προστασία του κλίματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε οικονομική ανάκαμψη και αύξηση όσον αφορά και την εξυγίανση του οικονομικού μας συστήματος. Στην Πολωνία έχουμε τους τρεις στόχους 20-20-20% και για την έρευνα, για την καθαρή τεχνολογία του άνθρακα, νέες τεχνολογίες, ε, για καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το κάνουμε αυτό και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη-μέλη το κάνουν αυτό από πλευρά τους, είναι πολύ σημαντικό και για την παιδεία εκπαίδευση ε, θα ήθελα να αναφέρω κάτι πολλά μπορούμε να πετύχουμε. Αν ξεκινήσουμε νωρί, ε, έγκαιρα, στο δημοτικό σχολείο, στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό και συνεχίσουμε μετά με μια προσέγγιση που θα ε, θέτει έμφαση στην γνώση και στην συνειδητοποίηση για τα περιβαλλοντικά προβλήματα, αυτό θα είναι η οδός προς το μέλλον. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια Βινιάλη από την Ιταλική Βουλή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μπροστά στην κρίση όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης ε, προετοιμάζουν ένα μείγμα ε, απαντήσεων έτσι ώστε να διατηρήσουν την απασχόληση, το εισόδημα, την ενίσχυση των επιχειρήσεων, επενδύσεις στην ενέργεια, κυρίως στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στο, για το περιβάλλον. Και όλα αυτά τα κάνουν λαμβάνοντα υπόψη δύο βασικά απαραίτητα στοιχεία. Το ένα είναι ότι θα πρέπει να, να διατηρήσουμε από τον έλεγχό μας την, τα δημόσια οικονομικά. Διότι εάν επιστρέψουμε σε εθνικιστικές πολιτικές θα είναι μια επιστροφή στο, στο παρελθόν. Το πρόβλημα είναι όχι να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, αλλά πώς πρέπει να το κάνουμε. Και αν θέλουμε μια άμεση απάντηση, θα πρέπει να αποδεσμεύσουμε τις, ενεργείες, τις των ατόμων και των επιχειρήσεων. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε ε, τις, ε, τις δυνατότητες που υπάρχουν. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τις ε, απαντήσεις ε, ε, που προσφέρουν οι επιχειρήσεις που μπορούν να δημιουργήσουν μια κοινωνία welfare και αυτό είναι το, θέμα, το πρώτο θέμα ε, στο οποίο παίζει ρόλο σημαντικό η επικουρικότητα. Λέμε πάρα πολύ σωστά ότι θα υπάρξει ανάκαμψη της οικονομίας εάν υπάρχει εμπιστοσύνη. Γι' αυτό θα πρέπει εμείς να ξεκινήσουμε να δείχνουμε εμπιστοσύνη στις πρωτοβουλίες των ατόμων και της κοινωνίας και των εταιριών. Θα πρέπει να δώσουμε αυτά παραδείγματα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, απλουστεύσουμε την γραφειοκρατία που αντιμετωπίζουν οι εταιρείε και οι σήμερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, απλουστεύσουμε τι διαδικασίε έτσι ώστε τα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσει να μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στα ε, οικονομικά πακέτα ε, ενίσχυσης ή στα στην, ενέργεια. Θα βγούμε από την κρίση μαζί σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει όμως να μπορέσουμε να παρεμβαίνουμε και μαζί και στα θέματα πολιτικής και στα θέματα της κοινωνίας. Ευχαριστώ. Ο, οποίος, ο επόμενος ομιλητής ο κ. Γκαλαζεύσκη από το ε, Κοινοβούλιο της Πολωνίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας ε, ακούσαμε πολλές φορές τον όρο προστατευτισμός. Ε, όλοι είπαν ότι πρόκειται για κάτι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Κανιά όμως αντιπροσωπεία δεν θέλει να παραδεχθεί ότι ο προστατευτισμός είναι ένας τρόπος για να ξεφύγει μια χώρα από την, από την κρίση. Και είναι μια επιλογή που κάνουν οι πολιτικοί. Και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Τοπολάνα και τον κύριο Μπαρόζο. Αυτό το φάντασμα, αν θέλετε, ε, ο τρόμος της, ε, του προστατευτισμού είναι τελείως θεωρητικός ή κάνουν κάτι τέτοιο συγκεκριμένα κράτη. Έχουμε παρεξηγήσει τις προθέσεις κάποιων Ευρωπαίων σε ηγετών ή ας πούμε τα μέτρα που υιοθέτησαν, που θέτησε η Αυστρία, ας πούμε, πέντε, η αυστρια ας πεντε χρονια μετα την προσχώρηση. Τι είναι και αυτά προστατευτισμός είναι. Και τέλο πάντων, τούτου λεχθέντο να τελειώσει και με μια νότα αισιοδοξία. Η κρίση μέχρι σε έναν βαθμό είναι καλά νέα διότι θα πρέπει όλοι να καθίσουμε και να σκεφτούμε είναι αποτελεσματικά αυτό τα οποία κάνουμε. Στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είχαμε ένα καλό παράδειγμα, το πακέτο για το κλίμα. Για άλλη μια φορά αξιολογήσαμε την προσέγγιση, ε, είδαμε και υπολογίσαμε το κόστος που συνεπάγει το πακέτο και καταλήξουμε σε κάποια συνένεση. Και αυτό ήταν μια καλή ένδειξη, διότι πρόκειται για ένα δύσκολο project και παρόλα αυτά υιοθετήθηκε μια υπεύθυνη στάση και λήφθησαν αποφάσεις. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής είναι η κυρία Άγκουας από, την, ε, από το Κοινοβούλιο της Πορτογαλίας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να εκφράσω την τιμή που αισθάνομαι ότι μπορώ να συμμετάσχω σε αυτή τη διάσκεψη για πρώτη φορά και θα ήθελα να προσθέσω σε αυτή τη συζήτηση που είναι τόσο σημαντική όσον αφορά την ανάκαμψη και την αντιμετώπιση της κρίσης να προσθέσω μια προοπτική που όπως εγώ μετριοπαθώς πιστεύω, πιστεύω ότι δεν πρέπει να αγνοηθεί. Και αυτή είναι η διάσταση που έχει αυτό το πρόβλημα και που έχει τα αίτια της στη οικονομική αυτή κρίση, οικονομική χρηματοπιστωτική κρίση, που είναι κρίση ηθικής, κρίση αξιών και αρχών, κρίση της ανθρώπινης φύσης, των ανθρώπων των ίδιων. Όταν ακούω εδώ όλους να αναφέρονται και σε όλες αυτές τις δύο μέρες να έχουμε αυτά τα κλειδιά, έννοιες κλειδιά, δηλαδή προσοχή όχι στον προστατευτισμό ας ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας και να είμαστε ενωμένοι γιατί αν ενωθούμε έτσι εμείς θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε την κρίση έχουμε ένα κοινωνικό πρότυπο που θα μας βοηθήσει και θα πρέπει να μπορέσουμε να το διατηρήσουμε Τώρα, όσον αφορά αυτά, αυτό που θέλω να ερωτήσω είναι το εξή. Μήπως η ίδια οικονομική ανάπτυξη που θέλουμε να πετύχουμε Εκείνο που είχαμε πιο πριν, πριν φτάσουμε σε αυτήν την κρίση, αυτό είναι που θέλουμε. Αυτή η οικονομική ανάπτυξη, η οικονομική ανάπτυξη τι σημαίνει. Θα είναι συνώνυμη της οικονομικής ανάπτυξης ε, όταν βλέπουμε ότι ε, με ένα τεράστιο ποσοστό που, ε, του παγκόσμιου πληθυσμού ζούμε κάτω από ένα δολάριο καθημερινά και όταν ζούμε σε μια οικονομία ξέφρενου καταναλωτισμού και όταν βλέπουμε ότι εδώ πάρα πολλοί άνθρωποι μένουν εκτός, αυτό είναι το ερώτημα το οποίο θέλω να θέσω. Τι θα κάνουμε με αυτό το πρόβλημα. Γιατί νομίζω ότι πρέπει ξεχωριστά να αντιμετωπιστεί αυτό μια νέα προσέγγιση κοινωνική που πρέπει να υιοθετήσουμε, μια νέα πολιτική προσέγγιση ως πολίτες, μια ευθύνη, υπευθυνότητα ατομική κάθε ενός από μας μπροστά στα κοινά προβλήματα που πρέπει να προσπαθήσουμε να τα αντιμετωπίσουμε από κοινού. Το σχολείο, η εκπαίδευση, η παιδεία είναι ο τόπος που πρέπει να ξεκινήσουμε. Και επίσης και την εντύπωση που θέλω να εκφράσω ότι όταν κάνουμε λόγο για το περιβάλλον και για το κλίμα χωρίς να έχουμε διασφαλίσει παγκόσμια να προσθέσουν όλες τις προσπάθειές τους υπέρ αυτής της προσπάθειας γιατί δεν θα είναι ε, αηφόρα αυτή η προσπάθεια αν μόνο ένα μέρος των πολιτών αυτού του πλανήτη ακολουθεί αυτούς τους στόχους. Πρέπει όλοι να τους ακολουθήσουμε. Η εξή ερώτηση στη συνέχεια για το ε, πρέπει να απορριφθεί ο προστατευτισμός όπως προαναφέρθηκε. Εγώ συμφωνώ. Συμφωνώ ότι ο προστατευτισμός ε, πάντα είναι μια πηγή πολλών κακών. Όμως κάποιοι προστατευτισμοί είναι θέματα που ανεχόμαστε στην Ευρώπη. Και ρωτώ, γιατί η Ευρώπη για παράδειγμα δεν προσθέτει και εκείνη την προσπάθειά της και δεν καθορίζει την χρήση ενός ε, ε, μιας ε, δυνατότητας που θα πρέπει να προσπαθήσει να βρει ε, την, ανεξάρτητη, θέση στον κόσμο σε σχέση με μονοπόλια και που κοστίζουν δισεκατομμύρια σε αυτή την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος αγορητής, ο κύριος Γιούγκ από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να πω ότι δεν συμμερίζομαι αυτό το οποίο αισθάνομαι, διαισθάνομαι, ε, αυτή την ότι υπάρχει μια αισιοδοξία στις συζητήσεις μας. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο συνάδελφος από την Αυστρία. Είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Ο κύριος Λούντ, ο οποίος είναι ένας αναγνωρισμένος οικονομολόγος, μας είπε ότι η κρίση αυτή θα είναι θα κρατήσει τρει φορέ περισσότερο και θα διαρκέσει τρεις φορές περισσότερο και θα είναι τρεις φορές πιο βαθιά από αυτά που έχουμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν. Άρα χρειαζόμαστε φιλόδοξα μέτρα για να απαντήσουμε σε αυτή την κρίση. Και τα μέτρα αυτά δεν τα βλέπω εγώ να υιοθετούνται. Βλέπω κάποια εθνικά σχέδια, κάποια προγράμματα, έτσι λίγο ε, σε ε, άτακτα και χωρίς ιδιαίτερο συντονισμό για την ε, κατανάλωση και μετά βλέπω μια πολύ ντροπαλή στάση από πλευράς της Κομισιόν, για να τη χαρακτηρίσω απλώς και μόνο έτσι. Όμω οι προκλήσει είναι τεράστιε τι οποίε αντιμετωπίζουμε. Βλέπουμε ότι κάθε μέρα να χάνονται θέσει απασχόληση, χιλιάδε θέσει απασχόληση. Και θα πρέπει να περιμένουμε τον Απρίλιο, τον Μάιο για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και μετά υπάρχουν και τα βραχυπρόθεσμα μέτρα, η ανόρθωση τη ζήτηση, όλα αυτά τα βραχυπρόθεσμα μέτρα, στρατηγική τη Λισαβόνα, να χρηματοδοτήσουμε την έρευνα, να χρηματοδοτήσουμε την ενεργειακή πολιτική, να, να, χρηματοδοτήσουμε υποδομέ, όλα αυτά πολύ καλά. Αλλά πώ θα τα κάνουμε όλα αυτά. Δεν το βλέπουμε να γίνεται. Εγώ δεν βλέπω πώς θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Και πιστεύω ότι είμαστε πάρα πολύ ντροπαλοί και άτολμοι και ε, θα πρέπει και έχουμε ε, εφαρμόσει εμείς οι ίδιοι τον, τον, ένα περιορισμό στον εαυτό μας για τον προπολογισμό του 1% κτλ. Όμως πέραν του προπολογισμού μπορούμε να βρούμε και άλλους πόρους π.χ. την αγορά των ευρωομολόγων. Γιατί να μην ξεκινήσουμε, γιατί να μην ζητήσουμε, να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε ε, κάποιο δανεισμό ε, στην, αγορά μέσω ομολόγων ή δεν ξέρω τέλος πάντων 800 δισεκατομμύρια, 1000 δισεκατομμύρια ευρώ για να χρηματοδοτήσουμε όλες αυτά τα μέτρα τα οποία θέλουμε να εφαρμόσουμε. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο φοβάμαι θα ε, προσκρούσουμε σε έναν τείχο και εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε άμεσα αυτή την τόσο βαθιά κρίση. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Κρίλ από την Τσεχία, από το Τσεχικό Κοινοβούλιο. Eh, Ευχαριστώ Πρόεδρε, Κυρίε και κύριοι. Κατά τη διάρκεια τη ε, συνάντησή μα, συζητούσαμε για την εξέβρεση λύσεων για την οικονομική κρίση. Κάναμε λόγο επίση για γοργή δραστηριοποίηση, επίγουσα δράση, βραχυπρόθεσμα. Όλα αυτά πολύ ωραία, αλλά α μην αγνοούμε τι μεσοπρόθεσμε και μακροπρόθεσμε λύσει και στόχου, Ένα πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να υλοποιήσουμε σωστά σωστά την στρατηγική της Λισαβόνας. Διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τους στόχους του 2010, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει πιο ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά σε παγκόσμια κλίμακα η πιο αποτελεσματική και ανταγωνιστική μονάδα. Το 2004 αναθεωρήθηκε η στρατηγική της Λισαβόνας και μπορούμε με σαφήνεια, με σαφή τρόπο να δούμε ότι αποτυγχάνει η στρατηγική της Λισαβόνας. Όχι μόνο χωλένουμε και πόρο απέχουμε πίσω από τη ΣΥΠΑ, αλλά υπάρχει νέος κίνδυνος οι νέες υπερδυνάμεις της ε, Ασίας να μας προσπεράσουν. Χωρίς την ε, νέα καινοτόμα τεχνολογία, χωρίς νέες τεχνολογίες εχμής δεν μπορούμε να επιβιώσουμε στην παγκοσμιοποιημένη αγορά. Και οι στόχοι του 2010 που πρέπει να επιτευχθούν, το 3% του ΑΕΠ που πρέπει να δίνεται για την έρευνα για τις επενδύσεις δεν θα επιτευχθεί. Ούτε καν κατά το ίμιση δεν θα ε, καλύψουμε την απόσταση που πρέπει να καλυφθεί νομίζω ότι μια κα, κακομελετημένη, κακώς σχεδιασμένη στρατηγική είναι μεγάλο ε, κακό, χειρότερο από το να μην έχουμε καν καλή, ε, κάποια στρατηγική. Και τι θα γίνει με τους στόχους αυτούς μετά το 2010 σε σχέση με τη στρατηγική της Σαββόνας, σε σχέση με το Συμβούλιο, ποιε απαντήσεις θα δοθούν για αυτή τη στρατηγική. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω την Προεδρία τώρα στον Πρόεδρο Πέτερινγκ, παρακαλώ. Äh, Πώς με εξέπληξε αυτό. Ε, ήταν ξαφνική αυτή η παράδοση σκητάλης της Προεδρίας. Σύμφωνα με το δικό μου πρόγραμμα είχε διαφορετική μορφή η εξέλιξη της συνεδρίασης, όμως και τα πρόβλεπτα πρέπει κανείς να αντιμετωπίσει. Θα ήθελα ο Προεδρεύων του Συμβουλίου, ο Προεδρεύων κύριος Τοπολάνεκ να μπορέσει να συνοψίσει και μετά ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κύριος Μπαρόζο. Παρακαλώ κύριε Προεδρεύοντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Τοπολάνεκ, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι πράγματι ευγνώμων, ευγνώμων για όλες αυτές τις ε, παρεμβάσεις ε, από πλευρά σας. Ο Πολωνός κύριος έχει δίκιο. Ο στασιμοπληθωρισμός είναι χειρότερος από τον αποπληθωρισμό. Και έτσι εδώ μια ύφεση είναι χειρότερη από μια συρρήκνωση και όλα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να αντιδράσουμε έγκαιρα και σωστά. Πρέπει να είμαστε συνετοί. Το να πιστεύουμε ότι εμείς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση μόνοι μας είναι ένας μύθος. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτός ο μύθος σε μια πραγματική οικονομία. Ανοησία είναι αυτό. Εμείς ε, βρισκόμαστε εδώ για να απαμβλύνουμε τις επιπτώσεις της κρίσης και για να αναλάβουμε μέτρα για να ανακάμψει η οικονομία στο μέλλον. Μέχρι σήμερα στην Τσεχική Δημοκρατία λάβαμε μέτρα του 1% περίπου ε, του ΑΕΠ μας ένα δις ευρώ, λίγο παραπάνω από ένα δις ευρώ για την αντιμετώπιση της κρίσης. Μεταξύ της σημερινής ημερομηνία ε, και μέχρι τα τέλη του έτους ε, περαιτέρω 2% του ΑΕΠ μας θα προσθεθούν ως κονδύλια. Είναι ένα πολύ σοβαρό πακέτο μέτρων. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί που θα διαθέσουμε αυτά τα, κονδύλια και ποιες επιπτώσεις πολλαπλασιαστικές μπορούν να ε, ε, επακολουθήσουν για την ανάπτυξη, την απασχόληση, την διατήρηση και βελτίωση, αύξηση της παραγωγικότητας για την Σύνοδο του Μαΐου. Η Σύνοδος αυτή του Μαΐου δεν θα επιλύσει το πρόβλημα της ανεργίας βέβαια. Υφίσταται όμως για να συζητήσουμε την αποτελεσματικότητα των μέτρων, μέτρων και εργαλείων που έχουμε υιοθετήσει και να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις ε, στην ανάπτυξη όλων αυτών. Ποιες είναι οι προοπτικές για το μέλλον, τι θα κάνουμε στο άμεσο μέλλον αν θα θα αλλάξουμε αυτά τα μέτρα, αν λειτουργούν σωστά και αν θα τα διατηρήσουμε αναλύωτα. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Και αυτά επειδή η ε, τα φορολογικά κίνητρα, τα εκτελεστικά διοικητικά μέτρα δεν θα πρέπει να διαιωνίζονται αν αποτυγχάνουν. Γι' αυτό η αναθεώρηση έχει πολύ σημαντικό χαρακτήρα. Πρέπει σε όλα τα επίπεδα να αποτιμήσουμε και να δούμε τι μπορεί να γίνει. Έχω ανησυχίες βέβαια για τις προσδοκίες των πολιτών σε σχέση με το πακέτο για τις κλιματικές αλλαγές δεδομένης αυτής της κρίσης. Πράσινες θέσεις απασχόλησης και πρασίνισμα των προσπαθειών. Το κατανοώ αυτό. Θέλουμε όμως και μέτρα τα οποία θα μειώσουν το κόστος για τις βιομηχανίες μας. Αν θέλουμε να επιλύσουμε τα προβλήματα αυτής της κρίσης λοιπόν, αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να προαγάγουμε τις επενδύσεις ε, στην εξοικονόμηση ενέργειας. Επενδύσεις σε προγράμματα και σχέδια που θα μειώσουν το βάρος το διοικητικό, την γραφειοκρατική επιβάρυνση των πολιτών. Η εφετινή κρίση για το φυσικό αέριο και η οικονομική συρρήκνωση και ύφεση θα δείξουν ως λιδία λίθος αν είμαστε σοβαροί στα όσα λέμε και θέλουμε να να πράξουμε ή όχι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για όλου του πολίτε ε, στα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούσαμε ότι είναι ηθική κρίση. Κρίση αρχών και αξιών. Συμφωνώ με αυτό απόλυτα. Η οικονομική ανάπτυξη είναι απλώ ένα μέτρο της ε, μέτρησης ε, του επίπεδου ζωής. Υπάρχουν επίσης θέματα ασφάλειας, προσπελασιμότητας, θέματα περιβάλλοντος, θέματα ανάπτυξης και παιδείας. Αν αποτύχουμε στην διασφάλιση οικονομικής ανάπτυξης, πολύ δύσκολα θα μπορέσουμε να πετύχουμε ανάπτυξη στους άλλους τομείς. Είμαι κατά του ξέφρενου, της χωρίς όρια αισιόδοξη προσέγγισης και απορρίπτω επίσης μια μη σε, οικονομική, σε οικονομικά θεμέλια, μια μη οικονομική προσέγγιση των πραγμάτων. Δεν είναι δυνατόν εμείς ως πολιτικοί να πιστεύουμε ότι θα μπορούμε να επιβάλλουμε κάποιες αρχές μας ή κάποιες δικές μας προτάσεις. Θα οξύναμε τα προβλήματα έτσι. Το πρόβλημα δεν είναι πόσα κονδύλια θα διατεθούν, ποια κίνητρα θα δοθούν και μόνο και τελεία και παύλα. Είναι πολύ πιο σύνθετο το ζήτημα. Θα έκρουα κόδωνα κινδύνου κατά του, ε, των προτάσεων νέων ομολόγων και νέων κονδυλίων ΕΣΑΗ e που θα πρέπει να διατίθενται γιατί θα έχουμε το μεγάλο πρόβλημα της αποπληρωμής του κρατικού χρέους. Αυτό θα αποσταθεροποιούσε την Ευρωζώνη. Θα διαλύαμε τα πάντα και θα συλλέγαμε τα θράψματα επί δεκαετίες. Πρέπει να πάψουμε να ομφαλοσκοπούμε με αυτόν τον τρόπο και να δραστηριοποιηθούμε σωστά. Αν υιοθετήσουμε μια μονοπλευρη, μόνοβε, μονομερή, δράση με μέτρα τα οποία δεν θα τονώσουν την εμπιστοσύνη θα επιδεινωθεί η κρίση. Εμείς βρισκόμαστε εδώ πάνω, εσείς εκεί και πρέπει να είμαστε σύνετοι με ευφυή τρόπο, να, ε, με σόφρονα τρόπο να μπορέσουμε με τα αναγκαία μέτρα να ε, οδηγήσουμε τους πολίτες στο να αποκατασταθεί το κλίμα εμπιστοσύνης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτούς. Πρόεδρος ε, Πέτερινγκ, σας ευχαριστώ κύριε Προεδρεύοντα το Πολάνεκ. Τρεις συνάδελφοι θα λάβουν στη συνέχεια για τον λόγο όπως τον έχουν ζητήσει, Όμω ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο θα παρέμβει πρώτα και μετά οι τρει συνάδελφοι. Παρακαλώ κύριε πρόεδρε τη Επιτροπή έχετε τον λόγο. Ε, Χάσω για το θέμα αυτό τη σοβαρότητα τη κρίση. Σημερίζομαι απόλυτα τις ανησυχίες που εξέφρασαν πολλοί από εσάς που αναφερθήκατε με απόλυτη ειλικρίνεια στο θέμα αυτό και συμμερίζομαι απόλυτα και τα αισθήματα, τα ανυπομονησία τα οποία τρέφεται. Σαν ερετός ε, εκπρόσωπος, ε, σαν ερετή εκπρόσωποι που είστε των πολιτών σας, της χώρας σας, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά την διάσταση που έχει πάρει η κρίση και τα νέα στοιχεία τα οποία τη χαρακτηρίζουν στις ε, εισαγωγικέ μου παρατηρήσεις ήμουν απόλυτα ειλικρινής και αντικειμενικός σας είπα ότι η κατάσταση μπορεί να χειροτερεύσει πριν ε, αρχίζει να καλυτερεύει. Αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση πάρα πολύ σοβαρή στην Ευρώπη και όχι μόνο στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο θα έλεγα. Στι Ηνωμένε Πολιτείε και στι αναδυόμενε αγορέ που θεωρούσαν ε, όταν ξεκίνησε η κρίση ότι ήταν προστατευμένε ε, από τα προβλήματα αυτά τα οποία γεννήθηκαν στι Ηνωμένε Πολιτείε είναι η πρώτη κρίση της εποχής της παγκοσμιοποίησης αυτή εδώ που μας αποδεικνύει ότι όλοι εξαρτώμεθα από τους υπολείπους και αν ε, μια κρίση θίξει το, την καρδιά του χρηματοδοτικού συστήματο ε, συστήματος στις ΗΠΑ παραδείγματος χάρη οι συνέπειες ε, θα είναι παγκόσμιες και είδαμε πώς επλήγει η παγκόσμια ζήτηση. Και όχι μόνο η παγκόσμια ζήτηση, αλλά και η εμπιστοσύνη. Είτε είναι εμπιστοσύνη των επενδυτών, είτε είναι εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Μόνο αυτή είναι μια πρωτόγνωρη κρίση την οποία αντιμετωπίζουμε. Και απέναντι σε αυτή την κρίση, τι κάνει η Ευρώπη. Καταρχάς πιστεύω ότι η Ευρώπη, αν λάβουμε υπόψη μας ότι είμαστε 27 ξεχωριστά διαφορετικά κράτη-μέλη, αντέδρασε καλά σε γενικές γραμμές. Δεν μπορούμε όπως ε, είπαν ορισμένοι, να κάνουμε την σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μία χώρα, εμείς είμαστε 27 χώρες. Τούτο ελευθέντος πήραμε και κάποια μέτρα πριν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι το project το οποίο υπέβαλε η Κομισιόν, το υπέβαλε η Κομισιόν τον Νοέμβριο και το Δεκέμβριο ε, υιοθετήσαμε το πρόγραμμα ανάκαμψης, το οποίο δεν μπορεί να είναι σαν και αυτό των, ε, της διότι εμείς είμαστε 27 χώρες, άλλες από αυτές ανήκουν στη ζώνη ευρώ, άλλες δεν ανήκουν, άλλες ε, βρίσκονται σε ύφεση, άλλες έχουν, ε, ε, παρουσιάζουν ανάπτυξη. Επομένως ε, υπάρχουν διάφορα μέτρα με ενίσχυση του ισοζυγίου πληρωμών, έχουμε την, ε, την χρηματοδότηση του χρέους κτλ. Επομένως ε, από πλευράς πολιτικής, από πλευράς πώληση είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε ένα κοινό πρόγραμμα το οποίο να αντιμετωπίζει 27 διαφορετικές καταστάσεις. Παρόλα αυτά όμως πιστεύω ότι το αποτέλεσμα ήταν καλό. Εφαρμόσαμε ένα πρόγραμμα το οποίο λαμβάνει υπόψη αυτές τις διαφορετικές πραγματικές Βέβαια, θα πρέπει τώρα να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στην εκτέλεση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι δεν μπορούμε κάθε μέρα να γεννάμε μια καινούργια ιδέα και κάτι τέτοιο δεν θα ήταν και χρήσιμο εξάλλου. Δεν θα πρέπει να προσθέσουμε στην δυσκολία της κρίσης ε, την, ε, το φόβο, αν θέλετε, των ε, ηγετών, των πολιτικών ηγετών. Αυτή είναι η κατάσταση, αυτή πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πήραμε μια απόφαση, θα πρέπει να ε, εφαρμόσουμε την απόφαση αυτή και δεν θα πρέπει να δημιουργούμε νέες, νέα προβλήματα διαιρώντα, ας πούμε την ενιαία αγορά, διότι αλλιώ θα είμαστε όλοι χαμένοι. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο πιστεύω ότι θα πρέπει η εκτέλεση των μέτρων να γίνεται με έναν να υπάρχει μια, μια βοήθεια στην εκτέλεση των μέτρων, να μην χάνουμε από, από τα μάτια μας και τα βραχυπρόθεσμα αλλά και τα μεσοπρόθεσμα μέτρα. Γι' αυτό θα πρέπει να βελτιώσουμε την ε, συνολική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και θα πρέπει να επενδύουμε σε τομείς που έχουν μέλλον, όπως είπανε πολλοί από εσά, γιατί εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλο δυναμικό δημιουργία θέσεων απασχόληση σε όσα έχουν να κάνουν με τις μελλοντικές πολιτικές, πολιτικές ενέργεια, βιώσιμη ενέργεια, καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος κτλ. Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο δυναμικό, θα πρέπει να το ε, ενισχύσουμε και δεν θα πρέπει τα βραχυπρόθεσμα μέτρα μας να έρχονται σε αντίθεση με τα μέσο ή μακρόπρόθεσμα μέτρα. Θα πρέπει να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς ε, μεταξύ μας ε, Κάποιος είπε από εσά ότι έχουμε 1% στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Όντως, έχει δίκιο. Την επόμενη φορά όμως θα, μπορούσαμε να, θα μπορούσατε να μας βοηθήσετε ζητώντας από τις χώρες σας, διότι οι χώρες ήταν αυτές που είπαν ότι δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε το 1%. Το θυμόσαστε αυτό. Ωραία. Θα μπορούσατε κι εσείς να μας βοηθήσετε. Στην Υπάρχει, υπήρχε ένας, ένας όμιλος, ένα κλαμπ την τελευταία φορά που έλεγε το μέγιστο πρέπει να είναι το 1%. Και τώρα ξαφνικά οι ίδιοι στρέφονται προ την Ευρώπη και ζητάνε την Ευρώπη να τα βρει τα χρήματα αυτά. Ε, δεν τα έχει η Ευρώπη τα χρήματα αυτά. Θα πρέπει να γίνει μια δημοσιονομική προσπάθεια σε εθνικό επίπεδο, που θα πρέπει να είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο με τι ΗΠΑ. διότι εμεί έχουμε και αυτό με τους Επομένως, αυτό το οποίο θα δαπανίσουμε, αυτά τα οποία θα δαπανίσουν τα κράτη-μέλη στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής, επειδή αυξήθηκε η ενεργεία παραδείγματος χάρη, θα είναι πολύ πιο σημαντικό από αυτό το οποίο δαπανούν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Επομένως πρέπει να είμαστε απόλυτα ρεαλιστές και να εξετάσουμε την, εξετάζοντας την κατάσταση. Είναι σοβαρή η κατάσταση, αλλά δεν θα πρέπει ούτε να είμαστε ε, ανεύθυνα αισιόδοξοι, ούτε να φτάσουμε σε αυτή τη μυρολατρεία ε, και την απεσιοδοξία στην Ευρώπη. Γιατί είχε πει, ο, πει ένας από τους ε, πατέρες της, ε, της Ευρώπης ότι δεν θα πρέπει να είμαστε ούτε αισιόδοξοι ούτε απεσιόδοξοι αλλά ρεαλιστές. Σας ευχαριστώ στα Πορτογαλικά Ομπριγάδο Πρόεδρε Μπαρόζο. Εξαιρετικό θα ήταν αυτό για να ολοκληρώσουμε, αλλά έχουμε ακόμα τρεις συναδέλφους που αναμένουν να παρέμβουν η κυρία Μαρία Οφέλια Μορέρο από την Πορτογαλία, από την Πορτογαλική Βουλή. Παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να χαιρετήσω ιδιαίτερα το συμπατριώτη μου που είναι μεγάλη τιμή και περηφάνεια για μας, τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κύριο Μπαρόζο. Χαιρετίζω μία ακόμα ευκαιρία συνάντηση κοινοβουλευτικών με ευρωκοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Αυτή τη φορά σε σχέση με την κρίση και τις επιπτώσεις και το ξεπέρασμα αυτών και τι μπορεί να γίνει σε σχέση με τις χώρες μας. Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της κρίσης με άλλα λόγια. Και πιο σημαντικό η δυνατότητα να μπορέσει να υπάρξει εδώ η δυνατότητα δραστηριοποίησης. Τι μπορούμε επιπλέον να κάνουμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο και στα εθνικά επίπεδα για να ξεπεράσουμε την κρίση. Σήμερα ο κύριος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μπαρόζο για άλλη μια φορά κατέδειξε μέρη αυτού του προγράμματο. Κάνουμε λόγο για λύσεις που έχουν εφαρμοστεί ήδη εν μέρη και πρέπει ακόμα να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο στο μέλλον και ιδιαίτερα όσον αφορά τον χρηματοοικονομικό τομέα. <clears throat> στην ομάδα, στην πρώτη ομάδα για τις χθεσινές διαβουλεύσεις, οι συζητήσεις επικεντρωνόντουσαν στις επιχειρήσεις, κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, όπου είναι σημαντικό θέμα η διάθεση πιστώσεων για να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν καλύτερα. Σήμερα έχουμε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση πλέον ότι είναι πιο σημαντικό για την αηφορία των οικονομιών και ιδιαίτερα για την οικονομία της Πορτογαλίας, της δικής μου χώρας, να υποστηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις περισσότερο από τις μεγάλες ε, επιχειρήσεις. Και αυτό για ε, εργαζόμενους. Υπάρχουν εκατομμύρια εργαζόμενοι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό να βοηθήσουμε αυτές σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Λιγότερο έγινε λόγος για λύσεις για τους ανθρώπους όμως και πώς θα αποφύγουμε την ρήξη των εθνικών συστημάτων όσον αφορά χιλιάδες ή εκατομμύρια κιόλας ανέργους και το βάρος που αυτό θα συνεπάγεται για τις οικονομίες μας. Στην Ευρώπη υπάρχουν σήμερα πολλές κοινωνικές εντάσεις μεταξύ εργαζομένων που, μεταξύ εκείνων που έχουν θέση απασχόλησης εργασία και εκείνων που δεν έχουν. Και σε εμά υπήρχε και κάποια, υπάρχει και ε, το θέμα που βλέπουμε και την ξενοφοβία στην, ε, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το θέμα δεν θα είναι το θέμα της φυλής αλλά το θέμα της εργασίας όμως, της θέσης απασχόλησης και εδώ θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Και τέλος δεν μιλήσαμε εδώ για ένα πρόγραμμα το οποίο θεωρώ ότι έχει τεράστια σημασία, τις διατλαντικές σχέσεις, σχέσεις μεταξύ ΕΕ και ΕΠΑ, ΕΕ, για τον ενεργειακό ανεφοδιασμό για παράδειγμα, που αυτό είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ε, πυλώνες ε, για τα κράτη μας. Συνεργασία με τις ΕΠΑ, ΕΕ, με το πρόγραμμα Ομπάμα που έχει ήδη εγκριθεί, στις διατλαντικές σχέσεις που πρέπει να είναι ε, σχέσεις θέσεις ε, θετικές για να μην χάνουμε και ευκαιρίες. Ε, πολύ μεγάλη ε, σημασία να έχουμε επαφές με το Κογκρέσο, τον ΗΠΑ και από πλευρά της Ευρωβουλής θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα τέτοιων επαφών μεταξύ των Εθνικών Βουλών και Κοινοβουλίων και του Κογκρέσου στις ΗΠΑ. Να έχουμε στενές σχέσεις. Δεν θα πρέπει ακόμα πιστεύετε να δημιουργηθεί μια κοινοβουλευτική συνέλευση διατλαντική που θα ασχολείται με αυτά τα θέματα αυτών των επαφών. Ευχαριστώ ε, Μάλιστα σας ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφε και τώρα έχουμε παρόλα αυτά ακόμα τρεις αγορητές. Δύο καταρχήν με το όνομα Στέφανο, Στέφανο Σοφιάνσκι και Στε, πρώτα Στέπαν Σοφιάνσκι από την Βουλγαρική Βουλή παρακαλώ. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Βρισκόμαστε εδώ για να ορίσουμε τι ρόλο έχουν να παίξουν τα Εθνικά Κοινοβουλία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον αγώνα όλων μας για να ξεπεράσουμε την κρίση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον ε, κύριο Πέτερινγκ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Τσεχική Δημοκρατία που έχει την Προεδρία και οργάνωση τη συνεδρίαση αυτή. Τι εργαλεία έχουμε στη διάθεσή μας στους εθνικούς προπολογισμού, του, τα ευρωπαϊκά κονδύλια και του, τα δάνεια. Αν Απροπιώ βέβαια τα πράγματα λίγο. Αν δούμε όμως τα εθνικά κονδύλια για την ανάκαμψη της ε, κρίσης πραγματικά βλέπουμε ότι υπάρχει ένας κάποιος ε, προστατευτισμός σε όλα τα εθνικά σχέδια. Ε. Ε, αυτό δεν πρέπει να φοβηθούμε να το πούμε. Από εκεί πέρα υπάρχουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την σταθεροποίηση ε, τα ευρωπαϊκά κονδυλιά που χρησιμοποιούνται για το συντονισμό και την κάποια εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μετά έχουμε και τις τράπεζες, την τραπεζική χρηματοδότηση οι οποίες δανείζουν ε, έναντι κάποιου τιμήματος βρισκόμαστε εδώ για να βρούμε μια λύση να ξεπεράσουμε την κρίση για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε θέσεις εργασίας για να μπορέσουμε να προλάβουμε ανεργία για τα θέματα αυτά εργασίας όλα τα κράτη-μέλη έχουν τις δικές τους εμπειρίες δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες αλλά ακόμη και στις ανεπτυγμένες χώρες ε, Υπάρχει ακόμη αρκετή δουλειά που πρέπει να γίνει. Α δούμε όμω κάποιους άλλου τομεί, Τον ενεργειακό τομέα χρειαζόμαστε μια σαφέστερη πολιτική και προστασία διότι δεν έχουμε φτιάξει τα εναλλακτικά σενάρια, τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας και ούτε η ηλιακή ούτε η αιωλική ενέργεια έχει προωθηθεί όσο θα θέλαμε και βλέπουμε ότι η Ιαπωνική αν θέλετε βιομηχανία έχει ουσιαστικά ε, εισβάλλει στην ε, Ευρώπη Ε, η οικολογία, η διαφοροποίηση ε, και η θέση εργασίας είναι πολύ σημαντική τομής και τέλος η γεωργία, ένας άλλος τεράστιος τομέας που πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα Εγώ σαν βούλγαρος πολίτης δεν τρομάζω με το ενδεχόμενο να υπάρχουν κανόνες ακόμη και για την κυβέρνησή μου. Προχωρώ στον επόμενο μιλητή, του κύριο Σέρναχ από το Bundesrat στην Αυστρία. Ευχαριστώ αγαπητοί κύριοι πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ο κύριος Λάρσον είπε ότι η κρίση αυτή θα είναι τρεις φορές πιο βαθιά και θα διαρκέσει τρεις φορές πιο πολύ από ό,τι ξέρουμε μέχρι τώρα. Και ο Πρωθυπουργός Τοπολάνε και ο Πρόεδρος Κομπισιών κ. Μπαρόζο ε, αναφέρθηκαν στα σημεία κλειδιά είπε ότι έχουμε ένα σύνδρομο αν θέλετε προβλημάτων στον οικονομικό ε, ε, εργασιακό και άλλους τομείς και έχουμε και στη γωνία το, το ενεργειακό πρόβλημα να κρύβεται είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε λοιπόν πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα μετά την κρίση. Τρεις σε τρία, τέσσερα χρόνια. Εγώ σας λέω ένα πράγμα, θα υπάρχουν τεράστια, τεράστιες τιμές στον ενεργειακό τομέα. Γι' αυτό χρειάζεται να προλάβουμε λίγο τα πράγματα. Η σχέση κεντρικής τοπικής κυβέρνησης ε, θα πρέπει να είναι τέτοια που να δώσει τη δυνατότητα και στην τοπική αυτοδιοίκηση να ασχοληθεί με την ενέργεια. Να δώσει την ευκαιρία στον κόσμο να πάρει κάποιες αποφάσεις. Έχουμε ε, με τις καινούργιες ενέργειες, με τις ανανεώσιμες ενέργειες θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε και θέσεις εργασίας και όσον αφορά την πυρηνική ενέργεια θα πρέπει να δούμε ότι τα πράγματα όπως τα φοβόμαστε από το παρελθόν έχουν ξεπεραστεί και τα, η πυρηνική ενέργεια είναι πολύ καλύτερη και δημιουργεί και θέσεις εργασίας. Νομίζω λοιπόν ότι ε, αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή να γίνεται και να σκέφτονται ορισμένοι ότι πρέπει να μειωθούν οι ε, επενδύσεις για τον τομέα της ενέργειας αυτό δεν μπορούσε να είναι κάτι μοναχά προσωρινό και βεβαίως επανέρχομαι σα πριν κλείσω ναι για την ελεύθερη κυκλοφορία στην αγορά εργασίας και όχι στον προστατευτισμό ευχαριστώ λέει ο πρόεδρος ο κύριος Ζαουρά έχει το λόγο τώρα πρόεδρε ευχαριστώ πριν από λίγο μίλησα σαν έκανα την παρουσίαση αν θέλετε της ομάδα 2 ε, ομάδας εργασίας 2 για τις κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης τώρα θα κάνω προσωπικές μου παρατηρήσεις συμφωνώ με, εκείνου που είπαν ότι μερικοί ίσω έχουν υποτιμήσει εδώ στην Ευρώπη το μέγεθο της κρίση και υπάρχουν και πολλά πράγματα τα οποία δεν τα βλέπουμε καθαρά και με, αυτή την έννοια ίσως η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι κατακαιρματισμένη. Στη Herald Tribune την περασμένη εβδομάδα έχει βγει και ένα άρθρο που επικρίνει την ε, ε, πολιτική ο Ομπάμα γιατί ο Ομπάμα λέει κάνει πράγματα τα οποία αντιμετωπίζουν τα χειρότερα βεβαίως αλλά δεν αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο μιας μακρόχρονης ε, ύφεσης στις, ε, ε, θεωρείτε λοιπόν ότι το πακέτο το αμερικανικό το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από το ευρωπαϊκό ίσως δεν είναι επαρκές για να ξεπεραστούν τα προβλήματα. Ο Κρούμπαν λέει στο άρθρο του ότι αν ε, δεν επενδύσουμε ε, για να για να ισορροπήσουμε αυτό το κακλημένο επίπεδο θα γλιστρήσουμε και θα πέσουμε όλοι προς τα κάτω αν πράγματι ε, υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο λυπάμαι αλλά και τα ευρωπαϊκά μέτρα δεν είναι επαρκή τα εθνικά σχέδια για την ανάκαμψη είναι πολύ μικρά ε, και δεν αντιμετωπίζουν τα βασικά προβλήματα και αυτό που είπε ο κύριος το Πολάνε δεν αρκεί δεν άκου, άκουσα τίποτα για, τις, για την κλιματική αλλαγή παραδείγματος χάρη ποια είναι η θέση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, συνάντηση των G20 ότι είμαστε όλοι στην ίδια κατάσταση αλλά όχι ακριβώς ε, τα πράγματα είναι σοβαρά αλλά όχι ακριβώς πρέπει να βρούμε τους τρόπους να ξεπεράσουμε τα πράγματα δεν ξέρουμε πως ακριβώς ακούσα να λέγεται και γίνεται και λόγος για τα ευρώ ευρωομόλογα οι Αμερικανοί δρούν εν πάση περιπτώσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο αλλά γιατί είναι μια χώρα ναι αλλά και εμείς θα μπορούσαμε να δράσουμε ενωμένοι αυτό θα έπρεπε να κάνουμε κύριε Πρόεδρε Ευχαριστώ πολύ και τώρα θα δώσω το λόγο στους Προέδρους Σομπότκα και Βολτσέκ για να εξάγουν τα συμπεράσματά τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι κατανοώ βέβαια ότι αναμένεται να συνοψίσω κάποια πράγματα συμπερασματικά. Ξεκινώντας θέλω να ευχαριστήσω βέβαια τον πρόεδρο Πέτεριν και όλους τους ευρωβουλευτές ε, διότι έγινε δυνατή η διεξαγωγή αυτής της συνεδρίασης μεταξύ Εθνικών Βουλών και Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τέτοιες συναντήσεις μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων και της Ευρωβουλής, ε, τέτοιες ε, διαβουλεύσεις έχουν κέρια σημασία Πέρσι, κατά την Άνοιξη, όταν προετοιμάζαμε μια τέτοια συνάντηση, είχαμε ένα άλλο θέμα υπόψη. Όμω η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έχει τέτοια σημασία, ώστε επιλέξαμε αυτό το θέμα για τις διαβουλεύσεις μας στη συνέχεια. Και όπω ακούσαμε από τον κύριο Πρωθυπουργό, τον Πολανέκα, τον Υπουργό Οικονομία ε, Παύλο Σέκ και τον ε, Πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριο Μπαρόζο και τον ε, Επίτροπο για τα Δημοσιονομικά κύριο Αλμούνια και τον κύριο Τρισέ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. έχοντα ακούσει όλε τι παρεμβάσει αυτέ, νομίζω έχουμε συναγάγει θετικά και σωστά συμπεράσματα. Είμαστε ευγνώμονε και για τι ομάδε εργασία για το έργο που επετέλεσαν και του θέλουμε να ευχαριστήσουμε και για τις περιλήψεις που δόθηκαν. Σε όλες τις παρουσιάσεις ακούσαμε με σαφήνεια ότι απορρίπτουμε με κάθε τρόπο την ιδέα προστατευτικών, υιοθέτηση προστατευτικών μέτρων και τον εθνικό, την εθνική οικονομική προσέγγιση με τέτοιου είδους μέτρα υπό οποιαδήποτε μορφή μπορούν να λάβουν τα εθνικά κοινοβούλια, στα κράτη-μέλη και στην Ευρωβουλή. Δουλειά μας είναι να συνεισφέρουμε με κάθε τρόπο, επομιζόμενοι τις ευθύνε μας, να συνεισφέρουμε για την επίλυση της κρίσης αυτής υπό το νομοθετικό, ε, τον χαρακτήρα των νομοθετικών ε, ε, δυνατοτήτων που έχουμε ανάληψης πρωτοβουλίας. Θα πρέπει να αναλάβουμε άμεσα γοργά ρόλο κατεπηγόντως να δράσουμε. Δεν πρέπει να αποδυναμωθούν ωστόσο όμως τα κριτήρια του Μαστρίχτ όσον αφορά το χρέος ε, και το ε, έλλειμμα. Και ως ε, πρόεδρος της Γερουσίας στην Τσεχία θέλω να ευχαριστήσω όλους για την δυνατότητα αυτής της διεξαγωγής, αυτής της διακοινοβουλευτικής συνάντησης. Ελπίζω ότι θα σας ξαναδούμε στις διάφορες συναντήσεις και εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί στην Πράγα. Και πάλι θα ήθελα να σας προσκαλέσω σε ένα κοκτέιλ, για ένα ποτό στην συνέχεια και ο κύριος Βότσεκ και εγώ έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στο κτίριο όπου θα παρασχεθεί. Σας ευχαριστούμε και ελπίζουμε να σας ξαναδούμε εκεί. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αξιότιμοι φιλοξενούμενοι, προσκεκλημένοι, η ε, βαθυμένη οικονομική κρίση και η διαφορετική αντίδραση από πλευράς των κρατών μελών στην ανάληψη πρωτοβουλειών για να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση μας έδωσαν υλικό για αυτές τις συζητήσεις, πολυσχηδείς συζητήσεις. Ενδιαφέρουσες ιδέες παρουσιάστηκαν σε αυτές τις συζητήσεις, ενδιαφέρουσες προτάσεις για την διέοδο, διέξοδο από αυτή την κρίση. Θα έχουμε και την συνάντηση των Προέδρων των Βουλών των Κρατών Μελών και ο κύριος Πέτερινγκ θα είναι παρόν, ο κύριος Μπαρόζο επίσης θα συμμετάσχει και θα είναι η κυριότερη ε, για το θέμα της Ευρώπης και της αντιμετώπισης της κρίσης ε, και τα εθνικά κοινοβούλια εμπλέκονται σε αυτό το πλαίσιο. Με ευχαρίστηση θα διαβιβάσω τους καρπούς αυτής της συνάντησης από τα εθνικά κοινοβούλια αυτής της συνάντησής μας στην ε, Σύνοδο των Παρισίων. Είναι κρίμα το ότι σε τέτοιες περιόδους και μάλιστα έκτη της κρίσης έχουμε τη δυνατότητα μόνο μιας τέτοιας συνάντησης σε σχέση με τις ευρωεκλογές μόνο μία διακοινοβουλευτική συνάντηση βλέπετε σε σχέση με την τσεχική προεδρία μας κατά τη διάρκεια της, του εξαμήνου μας. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα, όμως ελπίζουμε ότι οι επαφές μεταξύ Ευρωβουλής και των Εθνικών Κοινοβουλίων θα εμβαθυνθούν. Είναι ένας, μια αναγκαία συνάντηση και ε, εξυπηρετεί ε, τους πιο θετικούς στόχους. Και έτσι για τις επόμενες συζητήσεις ε, τις καλωσορίζουμε στα διάφορα επίπεδα οικονομική κρίση δεν είναι σαν την γρήπη την ε, εαρινή που μετά από κάποιες εβδομάδες μπορεί κανείς να την ξεπεράσει. Είμαι βέβαιος ότι θα ξανάρθουμε, θα επιστρέψουμε σε αυτά τα θέματα και θα τα ξανασυζητήσουμε στο εγγύς μέλλον. Υπό την Σουηδική Προεδρία για παράδειγμα και εύχομαι κάθε επιτυχία στην Σουηδική Προεδρία στο έργο που θα υπομειστεί. Ταυτόχρονα θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή σε αυτή τη συζήτηση, για το επικοδομητικό πνεύμα που δείξατε και ελπίζω ότι θα ξανασυναντηθούμε και θα ξανασυζητήσουμε και πάλι όταν ε, η Τσεχική Βουλή θα κάνει ένα δώρο στην Ευρωβουλή από πλευρά σας. Σας ευχαριστώ και πάλι Πρόεδρος Πέτερινγκ, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα ολοκληρώνοντας ε, να πω και εγώ δύο λόγια. Και με τρεις παρατηρήσεις να συνδυάσω ε, τα θέματα αυτά. Η κρίση στην οποία βρισκόμαστε είναι μια καινοφανής κρίση. Έχει διαφορετική μορφή από προηγούμενες, γι' αυτό δεν μπορεί να υπάρξει μια μαγική συνταγή. Το αποφασιστικό είναι από κοινού να δράσουμε όλοι μας τώρα και να βρούμε κοινέ απαντήσεις για αυτή την κρίση, για τον έλεγχο των τραπεζών του μέλλοντος. Και επ' αυτού θα πρέπει να σκεφτούμε κάποιες αρχές ε, τις οποίες θα τηρήσουμε. Η δική μας αρχή είναι η οικονομία της αγοράς, κοινωνική οικονομία της αγοράς. Είμαστε υπέρ της αγοράς, ταυτόχρονα αγορά αγορά πρέπει να υπηρετεί τους πολίτες. Γι' αυτό έχει ένα κοινωνικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίζει η αγορά. Και βρίσκεται και στη συνθήκη της Λισαβόνας η αρχή της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Σε αυτά τα ερωτήματα πρέπει να δώσουμε απαντήσεις. Το δεύτερο, το δεύτερο είναι ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο παρελθόν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα μέσα σε αυτή την εξέλιξη πετύχαμε πάρα πολλά πράγματα. Πετύχαμε την ολοκλήρωση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Όχι πλήρως και υπάρχουν κάποια θέματα που εκκρεμούν ακόμα και πρέπει να ολοκληρωθούν. Όμως έχουμε μια ελεύθερη κυκλοφορία και διακίνηση ατόμων, κεφαλαίων, υπηρεσιών και όποιος ξεκινά τώρα με προστατευτισμό, να κάνει λόγο για προστατευτισμό και προστατευτικά μέτρα σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση θα κατέστρεφε αυτή την ενιαία εσωτερική αγορά. Και έτσι στα θεμέλια τα οποία δημιουργήσαμε δεν θα είμαστε σε παγκόσμιο πλαίσιο ανταγωνιστικοί. Γι' αυτό πρέπει κάθετα να αντισταθούμε σε αυτόν τον προστατευτισμό και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προς τα έξω παγκόσμια. Και δεύτερη παρατήρησή μου αγαπητοί συνάδελφοι είναι ότι το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα αν δεν είχαμε αυτό το ευρωπαϊκό κοινό νόμισμα το ευρώ σήμερα, εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είμαστε σε πολύ μεγαλύτερες ε, αναταράξεις και προβλήματα. Και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας η σταθερότητα του ευρωπαϊκού νομίσματος του ευρώ να διασφαλιστεί. Δεν μπορούμε να περάσουμε να διολυστήσουμε σε μια νοοτροπία όλο και περισσότερα ελλείμματα και χρέη να δημιουργούμε και στο τέλος τέλος να υπονομευθεί αυτό το ενιαίο νόμισμα το ευρώ και να καταρρεύσει. Θα ξαναγυρίσαμε στα εθνικά νομίσματα και θα είχαμε τις Αντιπαραθέσει μεταξύ εθνικών νομισμάτων μεταξύ των κρατών μελών με ανατιμήσει, υποτιμήσει, και στο τέλο θα καταστρέφαμε και την ενιαία εσωτερική αγορά. Γι' αυτό για τη σταθερότητα και η εσωτερική αγορά ανήκουν στην ίδια τροχιά και πρέπει να διασφαλιστούν μέσω του ευρώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω στο τέλο, καταρχήν όλου του αγορητέ μα, Δύο βρίσκονται εδώ ακόμα. Ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής Ζωζέ Μανουέλ Ντουραν Μπαρόζο που πάντα είναι ένα εταίρο για μα, για την Ευρωβουλή. Ήταν και είναι. Και για τα εθνικά κοινοβούλια επίση. Ήταν πάντα στι συναντήσει μα παρόν και θέλω από καρδιά να τον ευχαριστήσω. Να τον ευχαριστήσω και για το πνεύμα συνεργασία που δείχνει από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εύχομαι ό,τι καλύτερο στον κύριο Μπαρόζο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσωπικά. Ο κύριο Ζωζέ Μανουέμ Ντουράν Μπαρόζο είναι πάντα παρόν και τον ευχαριστούμε προσωπικά και την Επιτροπή. Επίση, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Πρίτανη Λάρσον του Πανεπιστημίου Λούντ που εκπροσωπεί α το πω έτσι και ταυτόχρονα την επόμενη, την Σουηδική Προεδρία κατά κάποιο τρόπο. Σας ευχαριστούμε και εσάς που είσαστε παρόν. Ρητά και κατηγορηματικά ευχαριστώ όμως τους δύο συναδέλφους μου. Ξεχωριστά τους ευχαριστώ. Το πρωτόκολλο προβλέπει καταρχήν να παρέμβει ο πρόεδρος από πλευράς της ε, Γερουσίας η έκφραση ε, των ευχαριστειών ε, προς αυτόν για τη συνεργασία με την Ευρωβουλή. Ταυτόχρονα όμως και προς τον εκπρόσωπο πρόσωπο της ε, Βουλής ε, της Τσεχίας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για αυτή την με ε, συναδελφικό πνεύμα επικοδομητική συνεργασία. Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας ώστε η Τσεχική Προεδρία να στεφθεί με επιτυχία. Και εσείς μπορείτε να παρέμβετε ώστε απόψε στην Βουλή της Τσεχίας να διασφαλίσετε μεγάλη πλειοψηφία για τη συνθήκη της Λισαβόνας. Διότι και η συνθήκη της Λισαβόνας είναι ένα λιθαράκι, ένα μέσο, ένα εργαλείο να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση με επιτυχία επιτυχία και έτσι να περάσει προς τον 20ο αιώνα με επιτυχία. Στο τέλος ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες που συνεισέφεραν για την επιτυχία αυτής της εκδήλωσης και τους εξαιρετικούς λέει ο πρόεδρος διερμηνής μας και θα ξανασυναντηθούμε λοιπόν τώρα στην παρουσίαση και σας εύχομαι και επιστροφή, καλή επιστροφή στις πατρίδες σας που ανήκουν όλες στην Ευρωπαϊκή μας Ένωση. Υπό αυτό λοιπόν το πνεύμα σας ευχαριστώ θερμά και σας εύχομαι ό,τι το καλύτερο.